Καλησπέρα σας. Να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής σε μειωμένη σύνθεση, από ό,τι φαίνεται. Γιατί δεν βλέπω να έχουν έρθει συγγητές για κάποια θέματα. Να περάσουμε τώρα στην έγκριση της ημερησίας διάταξης. Όπως γνωρίζετε, σε σχέση με την πρώτη εκδοχή που εστάλει. Απλώς να σας πω ότι η Ολομέλεια έδωσε μία εντελή για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο σχετικά με το Ταμείο Αλίας και επομένως το σημείο 12 της ημερησίας διάταξης δεν θα το δούμε σήμερα καθώς ε, θα πρέπει να υπάρχει συμφωνία στην Ολομέλεια. Δεν υπάρχει άλλη τροποποίηση. Συμφωνείτε? Σημείο 2 έγκριση των πρακτικών της συνεδρίας 3 Οκτωβρίου. Αν κανείς δεν θέσει κάποια αντίρρηση κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, σήμερα θα εγκριθούν τα πρακτικά. Περνάμε στο τρίτο σημείο, ανακοινώσει του Προέδρου. Όπως σας είπα, ξέρετε ότι η Ολομέλη ανέκρινε το Ταμείο και με αυτή τη ψηφορία δόθηκε εντελή να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, προκειμένου να επιτευχθεί μια συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Και βάσει του άρθρου 70 του κανονισμού και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις διαπραγματευτική ομάδα θα αποτελείται από τον πρόεδρο της Επιτροπής ή από έναν αντιπρόεδρο, τον συγητή και τους σκιώδεις συγητές και το περιεχόμενο της διαπραγματευτικής εντολής βασίζεται στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της Ολομέλειας. Η πρώτη συνεδρίαση νομίζω ότι προβλέπεται για τις 7 Νοεμβρίου και όπως πάντα, θα σας ενημερώνουμε σε όλες τις συνεδριάσεις της Επιτροπής μας πώς προχωρούν οι διαπραγματεύσεις στους τριμερείς διαλόγους. Ερωτήσεις? Να συνεχίσουμε. Σημείο 4. Κοινή οργάνωση αγορών στον τομέα των προϊόντων αλίας και υδατοκαλλιέργειας. Σε πρώτη ανάγνωση εγκρίθηκε ε, το Σεπτέμβριο του 2012 η πρόταση και το Συμβούλιο υιοθέτησε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση στις 17 Οκτωβρίου. Ενέκρινε το Συμβούλιο τη Συμφωνία της 8ης Μαΐου 2013 μετά από τρεις συνεδριάσεις ε, τριμερούς διαλόγου και εμείς εγκρίναμε στις 18 Ιουνίου με 20 ψήφους υπέρ και μία κατά. Τώρα προβλέπεται η παρουσίαση της σύστασης για την ε, δεύτερη ανάγνωση του Κοινοβουλίου και να υπάρχει και μία προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών 5 Νοεμβρίου το μεσημέρι έχει διοριστεί αυτή η προθεσμία. Η παρουσίαση θα έπρεπε να γίνει από τον κύριο Στίφενσον που δεν είναι εδώ. Κυρία Ρόσπαχ, έχετε το λόγο. Συγγνώμη, δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Επομένως, να θέσουμε την προθεσμία 5 Νοεμβρίου το μεσημέρι και θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Ρόσπαχ. Παρακαλώ. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαιρετισμού από τον κύριο Στίβενσον που δυστυχώς ε, δεν μπορεί να παρευρεθεί στη σημερινή συνεδρίαση. Συστήνει όμω να παρπέμψουμε το θέμα για τη δεύτερη ανάγνωση. Θα ήθελε πάρα πολύ να προχωρήσει και να κλείσει το θέμα αυτό. Αυτό είναι το μήνυμα που μου ζήτησε να μεταφέρω. Ευχαριστώ. Bien, pues, cumplida la misión. Πολύ ωραία. Αποστολή εξετελέσθη. Σα ευχαριστώ. Θέλει κανεί το λόγο. Πάμε στο επόμενο σημείο τη ημερική διάταξη λοιπόν. η ελευτική πολιτική. Θα ίδια και εδώ, όπως και για την προηγούμενη έκθεση. Έχουμε θέτηση σε πρώτη ανάγνωση από την Ολομέλεια. Κρίθηκε η συμφωνία στις 17 Ιουνίου και εμείς το πράξαμε με 20 ψήφου υπέρ μία κατά και τώρα θα γίνει παρουσίαση για τη δεύτερη ανάγνωση με την ίδια προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών 5 Νοεμβρίου. Ούτε η κυρία Ρόντου στην εδώ. Κυρία Μιλάνα. Ε, συμμετέχει σε μια ψηφορία σε άλλη επιτροπή κυρία Ρόντουστ ε, και δεν μπορούσε να παρευρεθεί. Νομίζω ότι αυτή η έκθεση θα εγκριθεί έτσι ως έχει. Επομένως, ε, η σύσταση που δίνεται είναι να εγκριθεί σε πρώτη ανάγνωση και καθορίζεται μια σύντομη προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών. Ερωτήσεις, λέει ο Πρόεδρος. Συνεχίζουμε λοιπόν. Περνάμε στο έκτο σημείο ο δασμολογικές ποστός τη Ένωση για τις εισαγωγέ προϊόντων της τη Κανάριας νήσους. Αυτό είναι ένα θέμα για το οποίο είμαι αρμόδιος. Εγώ νομίζω ότι στην περασμένη φορά ήδη είχαμε τη δυνατότητα για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Και αν συμφωνείτε, τι να κάνουμε, νομίζω ότι δεν είναι επίμαχο το θέμα. Έτσι λοιπόν να μου δώσω απευθείας το λόγο. Δηλαδή, να επιβεβαιώσω όσα είχαμε ήδη πει. Πρόκειται για μια έκθεση όπου εδώ θέλουμε να επικυρώσουμε μια κατάσταση που ισχύει από το 1991. Τώρα μου αρέσει εμένα πάρα πολύ να μιλάω για τις ε, άκρως μας περιοχές, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται να σας εξηγήσω εδώ. Και πάλι, περί την όσο πρόκειται, όπως σας είπα, το 1991 εν μέρη οι καθολικά καταργήθηκαν οι δασμοί για τις αγωγές οσμών προϊόντων αλίας της Κανέρης Νήσου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελειώνει αυτή η περίοδος και θα σταματήσουν να ισχύουν μέτρα την 1η Πρώτου 2014. Αυτή είναι η πρόβλεψη και φυσικά με όλες τις ε, θετικές εκθέσεις των Ισπανικών αρχών για την εφαρμογή αυτή των δεσμολογικών ποσοστώσεων θα αιτιολογεί το γιατί καλύπτει τις ε, ανάγκες της εσωτερικής αγοράς της Κανάριας νήσους και αυτό που κάνει η έκθεση είναι να εγκρίνει να υπάρξει συνέχιση, παράταση των ίδιων δημοσιολογικών ποσοστώσεων να γίνει λοιπόν ανανέωση από την 1η 1η 2014 και να ισχύει για την περίοδο 2014-2020. Το συζητήσαμε αυτό στην περισμένη συνεδρία της Επιτροπής μας και απλώς θέλουμε να επικυρώσουμε αυτό το θέμα. Η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών θα είναι μέχρι τις 6 Νοεμβρίου για να ψηφίσουμε το Νοέμβριο στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια το Δεκέμβριο έτσι ώστε να προλάβουμε και την προθεσμία την 1η Ιανουαρίου 2014. Εγώ θα δώσω την, ε, το λόγο στην Κομισιόν, αν θέλει. Ο κύριος Δεπίπερ. Thank Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να προσθέσω πολλά, διότι μας εξηγήσατε το περιεχόμενο της ε, έκθεσης, το οποίο είναι απόλυτα σαφές. Ε, είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις, σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις, αλλά δεν είναι μία πρόταση που θα πρέπει να προκαλέσει πολλές συζητήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα κάποιος το λόγο. Κανείς. Πολύ ωραία. 6 Νοεμβρίου, λοιπόν, ε, προθεσμία κατάθεση τροπολογιών. Σας ευχαριστώ. Μακάρι να μην ε, έχουμε προβλήματα για καμία έκθεση. Πάμε στο σημείο 7. Κατάργηση του κανονισμού 827-2004 για την απαγόρευση τη αγωγή των μεγαλόφιλων του Ατλαντικού, καταγωγή Βολιβία, Καμπότζη, τη σημερινή Γουενέα Γεωργία και Σιέρα Λεόνη, του κανονισμού 1036-2001. Και η εισηγητή είναι ο κύριο Ρωμέβα. Τι θα κάνουμε σήμερα. Ο κύριος Ρωμέβα θα παρουσιάσει το σχέδιο τη έκθεση και θα τη δώσω αμέσω το λόγο. Παρακαλώ, ευχαριστώ. Νομίζω ότι και αυτό το σημείο είναι εύκολο γιατί ουσιαστικά ε, εδώ προτείνω το να γίνει δεκτή πρόταση της Κομισιόν ε, για ε, την έκθεση αυτή. Υπάρχουν κάποια σημεία βέβαια σε ό,τι αφορά τον ίδιο τον κανονισμό. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι προέρχεται ο κανόνας αυτός από το ICAT και μάλιστα από τη δεκαετία του 90 όταν η καταπολέμηση της παράνομης λαθρέας και τότε ε, ξεκινούσε και ήταν πολύ σημαντική. Εγώ νομίζω ότι συνεχίζει να είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε να επαγρυπνούμε για πάρα πολλά θέματα που έχουν να κάνουν με την παράνομη λαθρέα και αναρχελία κυρίως όταν μιλάμε για κάποια είδη πιο ευάλωτα και καθόπιν θα δούμε και την έκθεση για τον ερυθρό τόνο, όμως εγώ νομίζω ότι το παράδειγμα του μεγαλόφθαλμου είναι ένα από τα βασικά παραδείγματα. Η πρόταση που κάνουμε στην Επιτροπή είναι απλώς να δεκτούμε την πρόταση της Κομισιόν Δηλαδή στο να εγκριθεί αυτή η πρόταση παρέκκλησης και πάντοτε βέβαια θα έχουμε κατά νου την ανάγκη να επαγρυπνούμε για τα ζητήματα αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ρωμέβα. Από την Κομισιόν θέλει κάποιο το λόγο. Πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε. Ε, εξηγήθηκε πολύ καλά το θέμα αυτό. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την έκθεση που είναι πολύ σαφής. Ε, παραμένει το θέμα η καταπολέμηση της ε, αλίας πλά, έχουμε όμως καλύτερα εργαλεία. Γι' αυτό δεν είναι ανάγκη να διατηρήσουμε τα παλιά μας εργαλεία. Γι' αυτό προτείνουμε να καταργήσουμε αυτόν τον κανονισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κάποια παρέμβαση. Όχι. Ωραία. Προθεσμία καταθέσεις τροπολογιών στις 11 Νοεμβρίου το μεσημέρι. 11 Νοεμβρίου. Περνάμε στο επόμενο σημείο, το 8, Πολιτές, σχέδιο αποκατάσταση του τόνου, του ερυθρού τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο. Εδώ η συγητή είναι και πάλι ο κύριος Ρωμέβα και θα μας παρουσιάσει το σχέδιο έκθεση. Παρακαλώ. Εδώ έχουμε κάπως μεγαλύτερο περιεχόμενο. Σε σχέση με την έκθεση αυτή και την προηγούμενη υπάρχει κάτι σημαντικό να πω σε ό,τι αφορά τι τροπολογίες. Σε τρεις εβδομάδες θα πάμε στον ICAT, μια αντιπροσωπεία θα πάει στον ICAT και ίσως να υπάρχει κάποια τροποποίηση. Δεν έχει προβλεφθεί, αλλά είναι δυνατό. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκαθαρίσω ότι θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να μπορούμε να κάνουμε τροπολογίες μετά την επιστροφή μας ε, από το ICAT που θα γίνει στο κάμπο. Τώρα, εδώ απλώς εξηγούμε τους κανόνες που θετήθηκαν στο τελευταίο ICAT και δεν χρειάζεται να συζητήσουμε κάτι επί το περιεχομένου. Να υπενθυμίσω όμως ότι η συζήτηση που θα έχουμε και ίσως η Κομισιόν εδώ να μας δώσει τα φώτα της σε σχέση με τη γραμμή που θα υπερασπίσει βρίσκεται επιτάπητος και μια δυνατότητα που θα ζητήσουμε είναι να συζητήσουμε το θέμα του ΤΑΚ και τον Ερυθρό Τόνο το 2013. Δεν έχουμε καμία νέα αξιολόγηση που να αιτιολογεί αυτό το μέτρο και επομένως η Επιστημονική Επιτροπή ε, και εγώ συμφωνώ με την ανάλυση αυτή εφαρμόζει την αρχή της πρόληψης που λέει εφόσον δεν έχουμε στοιχεία αξιόπιστα που να δικαιολογούν την αύξηση των ΤΑΚ ε, τότε εμείς θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια πολιτική που να σέβεται τα κριτήρια που έχουμε θετήσει μέχρι τώρα και επιμένω ότι δεν υπάρχουν επιστημονικές αποδείξεις που να τη βελτίωση του αποθέματος. Έτσι λοιπόν εγώ νομίζω ότι πρέπει να διατηρήσουμε το κριτήριο της σοφροσύνης και σε ό,τι αφορά το θέμα της συνοχής με το κείμενο που έχουμε ήδη εγκρίνει για την κοινή πολιτική, όπου απαιτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια πολιτική που να βασίζεται στα επίπεδα που να είναι άνω της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης, έχουμε μία ευθύνη να διατηρήσουμε τη δυναμική αυτή. Τώρα, σε σχέση με τη συγκεκριμένη έκθεση, είχαμε εδώ τρία ζητήματα, πολύ συγκεκριμένα ζητείτε από το ICAT να αλλάξει, να τροποποιηθεί ε, η εποχή της Ελίας και τροποποιούνται οι κανόνες για τα ε, γρηγρή και για άλλα σκάφη, για τα σκάφη που με συρτή και αν υπάρχει κάποιο θέμα που εμείς προτείνουμε εδώ είναι μία διευκρίνηση, όχι μία τροποποίηση. Δεν αλλάζει το κείμενο, αλλά δεδομένου ότι η φράση σε μία από τις πτυχές ε, του κανονισμού ICAT είναι αμφίσιμη, δηλαδή γίνεται μία αναφορά κατά τη διάρκεια όλου του έτους ε, του ερθού τρόνου να επιτρέπεται και η με άλλα αλληλευτικά εργαλεία, αυτή η πρόταση, επειδή μας μπερδεύει, εγώ προτείνω να την διευκρινίσουμε. Και αυτή την πρόταση κάνω εδώ στην Επιτροπή Αλίας, να τροποποιήσουμε το κείμενο καθιστώντας πιο συγκεκριμένο το είδος των αλλιευτικών εργαλείων. Δηλαδή θα πρέπει να αναφερθούμε συγκεκριμένα στις διατάξεις παγίδευση τόνου, στην καθετή και στα μικρά παραγάδια. Προτείνω λοιπόν αυτή την τροποποίηση για να ξεκαθαρίσουμε το κείμενο. Δεν αλλάζει ουσιαστικά το νόημα και νομίζω ότι πρέπει να είναι αποδεκτή αυτή η τροπολογία. Και επιμένω ότι όταν γυρίσουμε από το ταξίδι μας το ΕΚΑΤ μπορεί να γίνει κάποια τροποποίηση που θα πρέπει να την έχουμε υπόψη. Όμως αυτό έχει να κάνει με το χρονοδιάγραμμα, θα το μπορούσαμε να το ξανασυζητήσουμε. Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Ρωμέβα από την πλευρά της Κομισιόν. So, um, yes, uh, Mr. Omeva raises uh, uh, Δύο ενδιαφέροντα σημεία. Νομίζω ότι το θέμα των ΤΑΚ, η συζήτηση συνεχίζεται και δεν μπορώ να ε, εκφέρω ακριβή σχόλια εκτός από αυτά του παρελθόντος που σχετίζονται ε, με την πρότασή μας να ευθυγραμμιστούμε με τις συστάσεις και για το εάν πρέπει ε, να αλλάξουμε την αποδοτικότητα ε, θα ήθελα να συζητήσω με τους ειδικού στο άνοιγμα του προγράμματος. Ευχαριστώ για τα σχόλια, αλλά για την ώρα δεν μπορώ να σας πω περισσότερα για το θέμα. Ευχαριστώ τον κύριο Ντεπίπερο, κύριος Μιλάνα. κάτι πολύ γρήγορα. Σε σχέση με τα ληφτικά εργαλεία. Εν μέρει μπορώ να συμφωνήσω με τα όσα είπατε Δηλαδή ότι πρέπει να γίνεται ελεία με πιο αλληλευτικά εργαλεία, ότι αυτό μπορεί να διευρυνθεί. Όμως από την άλλη μπορεί να έχουμε πρόβλημα ελέγχου για τα εργαλεία αυτά. Όμως εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Αν τελικά καταλήξουμε στην τροποποίηση του ποσοστού της ποσόστοσης αν θα έπρεπε να φτάσουμε εκεί. Εγώ νομίζω πρέπει να κάνουμε μία πρόταση για να κατανοήσουμε πώς ε, κατευθύνεται αυτή η αύξηση του ποσοστού και πώς συνδέεται με την χρήση πιο επιλεκτικών εργαλείων. Γιατί είναι σαφές αν τελικά η αύξηση της ποστόσωσης μπορεί να οδηγήσει στη χρήση πρακτικών ε, λιγότερο επιλεκτικών μεγάλης βιομηχανικής αλίας. Αυτό είναι πιο επώδυνο από το να χρησιμοποιήσουμε τα επιλεκτικά εργαλεία. Και αυτό το λέω γιατί σήμερα έχουμε πάρα πολύ μεγάλη παράνομη αλία ε, στον τόνο και προέρχεται ακριβώς από την απουσία ποσόστοσης. Και μάλιστα χρησιμοποιούνται και μέσα πολύ πιο επικίνδυνα, εργαλεία πολύ πιο επικίνδυνα. Επομένως, ε, κάτι έξυπνο που θα έπρεπε να κάνουμε είναι να έχουμε μία ποσόστοση που θα μπορούσε να μας χρησιμεύσει για την καταπολέμηση της παράνομης αλίας. Ευχαριστώ κυρία Φράγκα. Εγώ διάβασα την τροπολογία του κυρίου Ρωμέβα και δεν ξέρω αν προσφέρει κάτι σε σχέση με το αρχικό του κείμενο της Κομισιόν. Νομίζω ότι δεν συνεισφέρει αυτή η τροπολογία. Εγώ θα προτιμούσα το κείμενο της Κομισιόν που είναι πολύ πιο γενικό. Και δεν βλέπω την αναγκαιότητα για αυτή την τροπολογία. Θα ήθελα να ακούσω και ποια είναι η άποψη της Κομισιόν, αν είναι υπέρ αυτής της τροπολογίας ή, προτι... ή προτιμά το αρχικό κείμενο. Εγώ προτιμά το αρχικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα για τα ΤΑΚ και τις ποσοστώσεις σας τα αφήσουμε για μετά τη συνεδρίαση με το ICAT. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Φράγα. Κομισιόν, θέλετε να απαντήσετε στην ερώτηση της κυρίας Φράγα να μας πείτε ποια είναι η άποψή σας. Ε, προτιμάτε την τροπολογία ή το κείμενό σας, κύριε Τεπίπερ. Νομίζω ότι θα διατηρήσουμε τη θέση μας και την πρότασή μας. Μάλιστα, κύριε Ρωμέδα. Για το σχόλιο του συνάδελφου Μιλάνα. Είναι ανοιχτό το θέμα, είναι ένα θέμα που θα συζητήσουμε στο ICAT. Επομένω θα δούμε τι συμβαίνει. Εγώ κατάλαβα ότι έχουμε και το θέμα όχι μόνο της αύξηση, αλλά και της κατανομής της προσώστοσης και φυσικά αυτό θα είναι ένα από τα πιο καυτά θέματα της συζήτηση. Τώρα, η τροπολογία, κοιτάξτε, για να ξεκαθαρίσω το κείμενο το έκανα, για να μην είναι αμφίσιμο διευκρινίζω αυτά τα τρία είδη αλληλευτικών εργαλείων. Δεν είναι πολύ σχετική αυτή η τροπολογία. Αν θέλετε μπορούμε να το ξανασυζητήσουμε πριν την τελική ψηφοφορία. Μάλιστα, σχέση με την προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει και δυνατότητα, όπως είπε ο κ. Ρωμέβα, να συμπεριλάβουμε κάτι μετά τη συνεδρία του ΑΕΚΑΤ. Όμως δεν θα έχουμε χρόνο για να έχουμε μεταφράσεις και να πάμε στην Επιτροπή 16 και 17 Δεκεμβρίου. Έτσι λοιπόν διατηρούμε την προθεσμία της 11ης Νοεμβρίου και αν γίνει κάτι μετά τη συνεδρίαση του ΆΙΚΑ, υπάρχει κάποια τροπολογία, θα τις μετατρέψουμε σε προφορικές τροπολογίες και θα καταλήξουμε στη συμφωνία. Διαφορετικά δεν προλαβαίνουμε. Μου λένε ότι η καταληκτική προθεσμία για τη μετάφραση θα ήταν 21 Νοεμβρίου. Δεν θα έχουμε επιστρέψει από τον ΑΕΚΑΤ, δεν θα έχουμε τα τελικά αποτελέσματα. Α παραμείνει λοιπόν η προθεσμία στι 11 και αν υπάρχουν καινοτομίε θα δούμε τι θα κάνουμε με προφορικέ τροπολογίε ή θα επιλέξουμε κάποιο άλλο τρόπο. Ωραία. μικροφώνου, Πρόεδρος. Σημείο 9. Τροποποίηση ορισμένων κανονισμών στον τομέα τη αλληλεία και τη υγεία των ζώων λόγω τη αλλαγής του καθεστώ τη Μαγιότ έναντι τη Ένωση. Το θέμα αυτό το έχει αναλάβει ο κ. Φεραίρα, είναι ο εισηγητή. Ξέρετε την πλευρά του Συμβουλίου ζητήθηκε μια αλλαγή της νομικής βάσης για το άρθρο 43.2 της συνθήκης με απλή διαδικασία και στην προηγούμενη ολομέλη 22 Οκτωβρίου απορρίφθηκε το έκτακτο που είχε ζητήσει το Συμβούλιο. Επομένως υπάρχει ένα συμβιβασμός δηλαδή να κάνουμε την δυνατά μα να μπορεί να εφαρμοστεί αυτό το καθεστώς από τον Ιανουάριο του 2014 και σήμερα θα έχαμε την παρουσίαση του κυρίου Φερέιρα, όμως δεν ξέρω αν κάποιος έχει αναλάβει την παρουσίαση της έκθεσης αυτής, μάλιστα δεν σας είδα. Θα σας δώσω το λόγο για να την αντικαταστήσετε τον κύριο Φερέιρα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ ε, που με δεχθήκατε εδώ στην Επιτροπή σας, στην Επιτροπή Αλίας. Είμαι εδώ για να παρουσιάσω την ε, έκθεση του συναδέλφου ε, κυρίου Ζωάο Φερέιρα που μου ζήτησε να παρουσιάσω τα γενικά σημεία της έκθεσής του. Εξετάσατε μια πρώτη φορά τους κανονισμούς που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα υπενθυμίσω σύντομα τα βασικά σημεία του κανονισμού αυτού Πρώτα απ' όλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προτείνει ε, να μην ε, τα σειρώμενα δίχτυα να μην να απαγορεύονται ούτω ώστε να διαφυλαχθεί ο χώρος γύρω από το νησί Μαγιότ. Το δεύτερο πράγμα που προτείνεται και είναι σημαντικό είναι να δοθεί μια προθεσμία, ούτως ώστε να προσαρμοστεί στο κεκτημένο κυρίως όσον αφορά τις υποχρεώσεις σχετικά με την καταχώρηση και τον έλεγχο στον τομέα της αλληλείας, εφόσον υπάρχουν διάφορα σημεία γύρω από το νησί που δεν σχετίζονται με ειδικό τύπο εκφόρτωσης. Το τρίτο θέμα που είναι η υγεία των ζώων, όπου προτείνεται να δοθεί ε, στην Γαλλία ε, μία μεταβατική περίοδος όσον αφορά την Μαγιότ, ούτω ώστε να υπάρξουν όλες οι απαιτούμενες υποδομές για την απογραφή, ε, για την μεταφορά, για τον χειρισμό. Το αναφέρατε, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει μια συζήτηση σχετικά με τη νομική βάση του κανονισμού. Και χαίρομαι με τον Ζωάο για τη θέση της Επιτροπής Αλληλείας και προτείνουμε μια διπλή βάση, δηλαδή το άρθρο 349 να προσθεθεί στην νομική βάση που προτείνεται, που είχε προταθεί αρχικά σχετικά με το πρώτο σημείο του κανονισμού, δηλαδή τις προθεσμίες για τις ε, διάφορες ε, προτείνει να προσθεθεί ένα έτος ο εισηγητής ούτως ώστε να μπορέσει και η ηθαγενείς και η γαλλική δίκηση να θεσπίσουν κανονισμούς για την νιολόγηση και την καταχώρηση ε, των πλοίων. Όλοι πρέπει να ξέρουμε ότι την 1η Ιανουαρίου θα αλλάξει καθεστώς η γενουαριου θα αλλαξει Υπάρχει επίσης μια συζήτηση σχετικά ε, με την προστασία την ε, θαλάσσια και την απαγόρευση των γρηγρή θα πρέπει πρώτα απ' όλα να θεωρήσουμε ότι είναι το μεγαλύτερο ε, θαλάσσιο πάρκο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται εκεί και η κατάστασή του στον Ινδικό ωκεανό το κάνει ένα φυσικό ε, πάρκο πάρα πολύ μεγάλης ε, ομορφιάς και υπάρχει μεγάλη βιοπικιλότητα, μοναδική βιοπικιλότητα. Αυτό το πάρκο, το φυσικό της Μαγιότ καλύπτει 1100 τετραγωνικά χιλιόμετρα, 185 ε, υφάλους και 281 χιλιόμετρα ε, ακτές ε, και κοράλια που έχουν ε, καταχωριστεί. Θα πρέπει επίσης οι κοραλιογενείς ύφαλοι να προστατευθούν. Έχουμε mangrove 303.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και πάρα πολλά είδη με 750 είδη ε, ψαριών ε, θηλαστικά δηλαδή το εντέταρτο τέταρτο της παγκόσμιας βιοπικιλότητας, την μόνιμη παρουσία επίσης χελωνών και πάρα πολλοί ε, τύποι ε, οφορίας και αναπαραγωγής. Θα πρέπει λοιπόν να προστατευτεί η θαλάσσια βιοπικιλότητα που υπάρχει εκεί. Νομίζω λοιπόν ότι η Επιτροπή θα πρέπει να προστατεύσει αυτήν την εξαιρετική κληρονομιά δίδοντας στους ε, Μαόρε ε, αλληλείς τις δυνατότητες να επιτύχουν, να αναπτυχθούν και εκεί έχουμε τις κατευθυντήριες γραμμές αυτού του κανονισμού. Το σύνολο των αλλιευτικών πλοίων ε, και τα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης του Φυσικού Πάρκου της Μαγιώτα θα μπορούν να καθοδηγούνται από αυτήν την λεπτομερή ενδελεχή έκθεση για την οποία όλοι συμφωνούμε για να προ... προστατευτεί η λίμνο θάλασσα. Θα πρέπει τα πλοία ε, με σημαία ε, της Μαγιότ ε, να είναι πέραν των 24 ναυτικών μιλίων που είναι τα όρια της ζώνης θα πρέπει ε, τα, τα μεγάλα πλοία με ε, να μπορούν να λιεύσουν εκτός της ζώνης αυτούς, αυτά τα ψάρια και για, και για να είναι αυτό δυνατό ε, θα πρέπει τα πλοία μέχρι άνω των 12 μέτρων δεν θα μπορούν να ψαρεύουν στο φυσικό πάρκο της Μαγιώτα ε, που βρίσκεται στην αποκλειστική οικονομική ζώνη. Και αυτή είναι η θέση την οποία υποστηρίζει ο εισηγητής. Αν δεν υπάρχει αυτή η αγγίηση ε, για τους αλληλείς που θα πρέπει να ε, αλλιεύουν, όχι για εξαγωγή, αλλά για να μπορούν οι ίδιοι να καταναλώνουν τα ψάρια αυτά και για να έχουν ένα τρόφιμο το οποίο είναι ουσιαστικό για τον πληθυσμό που είναι ακόμα πάρα πολύ φτωχό. Ο πληθυσμό με τον Επίτροπο Χαν πήγαμε ε, στην ε, Μαγιότ, αλλά νομίζω ότι όλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει ποια είναι η κατάσταση στην περιοχή Νομίζω λοιπόν ότι η μικρή αλληλεία θα πρέπει να έχει δυνατότητα και να μην βρίσκεται ε, σε περίπτωση όπου δεν θα μπορεί ε, να αλλιεύει πέραν των 24 ναυτικών μιλίων. Ε, η, υδατοκαλλιέργεια και η αλληλεία παρόλο που η δατοκαλλιέργεια δεν περιλαμβάνεται στην εισήγηση, προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες για την ανάπτυξη του νησιού αυτού, εάν εφόσον βεβαίως προσανατολίσουμε εφ' τα μέτρα προς μια καλή κατεύθυνση, δηλαδή ε, την προστασία της λιμνοθάλασσης, την προστασία των κοραλιογενών υφάλων και δυνατότητα για τους αλληλείς να ψαρεύουν υπέρ του τοπικού πληθυσμού και όχι για εξαγωγή. Ευχαριστούμε. Καταρχήν να δώσουμε το λόγο στην Κομισιόν. Ο κύριος Τεπίπερ. Um, we, have to take note because, uh, Ναι, θα πρέπει να σημειώσω αυτά που άκουσα, διότι ο εμπειρογνώμονάς μου δεν είναι παρόν, δεν μπορώ να απαντήσω, απλά σημειώνω. Φράγα. Κυρία Φράγα. Εγώ διαβάζα πολύ προσεκτικά την έκθεση αυτή. Και έχω κάποια προβλήματα με το να αναβάλουμε τις ημερομηνίες. Εγώ νομίζω ότι για να γίνει μια καταχώρηση που θα πρέπει ήδη να λειτουργεί και υπάρχει εδώ και μια προθεσμία δύο χρόνια δηλαδή να επεκτείνουμε και την προθεσμία αυτή για την ιολόγηση νομίζω ότι είναι υπερβολικό. Αν κάποιος ε, δεν μου αποδείξει ότι αιτιολογείται όντως, εγώ δεν θα ήμουν υπέρ. Και σε σχέση για το φυσικό θαλάσσιο πάρκο της Μαγιότ. Γιατί αν διαβάσει κάποιος εδώ την αιτιολογική έκθεση, πίσω από όλα αυτά βρίσκεται η πρόθεση, τα μεγάλα γρηγρή που αλλιεύουν ε, στη ζώνη αυτή ε, να διευρυνθούν ε, δηλαδή τα μίλια που υπάρχουν που ήδη είναι πάνω από 100 Γίνεται λοιπόν ε, να γίνεται η προσπάθεια τα μίλια αυτά από 100 να γίνουν 200 για την παρέκκληση και διάβασα την έκθεση. Ε, λέγεται ότι η Ελία γρήγορη έχει αρνητικό εντύπωση για το θαλάσσιο πάρκο της Μαγιώτε και τα λοιπά και δεν ξέρουμε αν ελεύουν εκεί. Κάτι που είναι ψεύτικο γιατί όλα τα μεγάλα σκάφη που αλλιεύουν και όλα τα γρηγροί έχουν άδεια και το επιβεβαίωσε η Μαγιώτα αυτό, γι' αυτό δεν καταλαβαίνω πολύ καλά ούτε καν ε, την αιτιολόγηση που δίνεται εδώ. Και όπως ξέρετε, όλα μιλάμε για ιδιαίτερα μεταναστευτικά είδη, για εξόχως μεταναστευτικά είδη και το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να τα κλείσουμε αυτά τα ψάρια σε μία ζώνη. Επομένως, ε, το, δεν μπορούμε να κλείνουμε τις ε, ζώνες και να απαγορεύουμε την ελίκη, αλλά πρέπει να ελέγχουμε περισσότερο την ελιευτική προσπάθεια. Εγώ λοιπόν ε, δεν συμφωνώ με αυτή την πρόταση που γίνεται και νομίζω ότι εδώ γίνεται μία προσπάθεια να διευρυθούν τα μίλια της παρέκκλησης για την ελεύθερη πρόσβαση. Εγώ δεν είμαι υπέρ λοιπόν των όσων λέγονται εδώ. Θέλω να πω ότι δεν αιτιολογούνται οι παρατηρήσεις του εισηγητή στην έκθεσή του. Ουσιαστικά απευθύνονται στη βιομηχανική ελεία και στην ελεία του τόνου και εγώ επιμένω ότι εδώ μιλάμε για εξόχως μεταναστευτικά είδη, πρέπει να τα μεταχειριστούμε διαφορετικά. Και καθώς η ζώνη αυτή ουσιαστικά ρυθμίζεται από κάποιους κανόνες ε, που ισχύουν για την ε, περιοχή και αυτό είναι ένας επιπλέον λόγος που με κάνει να διαφωνώ με την πρόταση του εισηγητή. Ευχαριστώ κυρία Λοβίν. Ε, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Φυσικά, λυπάμαι που δεν είναι παρόν ο εισηγητής. Ε, πάντως ευχαριστώ για την εξήγηση της έκθεσης αυτής. Επίσης, λυπάμαι ακόμα περισσότερο που δεν είναι εδώ παρόν ο εμπειρογνώμων της Κομισιόν για να απαντήσει σε ερωτήσεις. Είναι σχεδόν σπατάλη δυνάμεων να κάνουμε οποιαδήποτε δήλωση ή ερώτηση. Πάντως θα θέσω τις ερωτήσεις, μας, τις ερωτήσεις μου και θα περιμένω μήπως εμφανιστεί απάντηση με κάποιο τρόπο. Οι ερωτήσεις λοιπόν αφορούν κυρίως ε, το φυσικό πάρκο της Μαγιότ. Εγώ δεν βλέπω στην έκθεση αυτή κανέναν σχετικό ορισμό. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω τι διαφορά έχει από τα 24 ναυτικά μίλια. Από τη ζώνη 24, 24 ε, μιλίων που, υπάρχουν στην αρχική πρόταση, που υπάρχει στην αρχική πρόταση. Επίσης, συμφωνώ με την κυρία Φράγκα σχετικά με την παράταση της προθεσμίας Συμφωνώ μάλλον ότι η παράταση της προθεσμίας ε, για ε, την καταγραφή του στόλου φαίνεται τελείως ακατάλληλο μέτρο, δεν ενδείκνεται. Και θα ήθελα επίσης ε, σε ε, σχετικά ε, σχέδιο ανάπτυξης που έχει υποβάλει η Γαλλία στην IOTC και πώς αυτό θα αυξήσει το δυναμικό στην περιοχή. Δεν νομίζω απαραίτητα ότι είμαστε υπέρ μιας απεριόριστης αύξησης του αλληλευτικού δυναμικού στον Ινδικό ωκεανό. Δεν είναι κάτι λοιπόν που θέλουμε να στηρίξουμε. Όσον αφορά αυτά που είπε η κυρία Φράγα σχετικά με τα γρηγρή και τον τόνο, Νομίζω ότι τα σκάφη αυτά εντός των προστατευομένων περιοχών ε, δεν ε, αλλιεύουν μόνο τόνο. Νομίζω ότι έχουν και παρεπίπτωτα αλλιεύματα όπως είναι ε, οι θαλάσσιες χελώνες ή οι καρχαρίες. Μπορεί λοιπόν να ε, είναι λογικό να απαγορεύσουμε τα σκάφη αυτά εντός μιας προστατευόμενης περιοχής. Και επίσης όσον αφορά το επίμαχο ζήτημα της νομικής βάσης, νομίζω ότι το μεγαλύτερο μέρος του Κοινοβουλίου συμφωνεί να μην επιτρέψουμε στο Συμβούλιο να μπορεί να τροποποιεί κανονισμούς χωρίς τη διαδικασία της συναπόφασης. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, άλλη παρέμβαση. Κύριε Τόμας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω για τους συναδέλφους που θέλουν λεπτομέρειες για το θαλάσσιο πάρκο, για να δούνε για τις ζώνες αυτές, την διαμόρφωση ζωνών προστατευομένων, πρέπει να ζητηθούν λεπτομέρειες για το τι είναι αυτό το θαλάσσιο πάρκο ε, του Μαγιότ, πώς έχει διαμορφωθεί, ποια είναι τα θαλάσσια τροτά οικοσυστήματα, ποιες είναι οι προτεραιότητες περιβαλλοντικής προστασίας, ούτω ώστε να έχουμε μια ιδέα γιατί ο εισηγητής προτείνει το μέτρο αυτό που δεν είναι να κλείσει μια αλλιευτική ζώνη, θα πρέπει βεβαίω αυτό να το ελέγξουμε, αλλά να ε, προσαρμόσουμε την αλληλεία ανάλογα με την προστασία που απαιτείται για αυτό το πάρκο. Να επιτρέπεται σε ορισμένες ζώνες. Θα πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας την πράξη αυτή που δίνει τον ορισμό του θαλασσίου πάρκου ε, του Μαγιότ στη Γαλλία η Επιτροπή Διαχείρισης του Θαλασσίου Πάρκου αποτελείται από ένα μέρος εθνικών γαλλικών αρχών και ένα μέρος τοπικών αρχών ε, ένα μέρος κυβερνητικό, ένα μέρος ειδικών. Έχει λοιπόν μια διακυβέρνηση η οποία είναι πολύ στενής, πολυκλαδική και θα πρέπει να έχουμε τα επιχειρήματα, χρειαζόμαστε τα έγγραφα αυτά για να έχουμε μια ιδέα. Θα πρέπει λοιπόν ο εισηγητής να μας υποβάλει τα κείμενα αυτά ως προς τις προθεσμίες ή την αναβολή υπάρχουν πολλοί περιορισμοί διοικητικοί από την αλλαγή του καθεστώτος με ελέγχους θα πρέπει να δούμε τι χρειάζεται ένας χρόνος παραπάνω, δύο χρόνια περισσότερο. Η ε, Κάρμεν πρεπει να δουμε τι χρειαζεται ενας χρονος παραπανω δυο χρονια περισσοτερο καρμεν φραγκα ζήτησε, ποιοι είναι οι λόγοι, θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη δίκηση όχι μόνο για την αλληλεία με βάση το νέο καθεστώς της μαγιότερα, να μην περιοριστούμε και στην αλληλεία και να δούμε τι πρέπει να γίνει γενικά για να μπορούμε να προσεγγίσουμε καλύτερα το θέμα. Ευχαριστώ κύριε Τόμας. κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε μερικά σημεία τα οποία αναφέρθηκαν. Ήδη ε, η κυρία Πίντης εν μέρη σε ορισμένα από τα ερωτήματα που τέθηκαν. Η Μαγιότ μέχρι σήμερα ήταν μέσα στο καθεστώς ε, των υπερποντίων εδαφών ε, και ε, είχε το καθεστώς ΦΕΔ. Το γεγονός ότι η Μαγιότ γίνεται περιφέρεια ευρωπαϊκή, ευρω... γίνεται Ευρώπη, είναι μια επανάσταση για αυτό το έδαφος που θα πρέπει να αναλάβει τις υποχρεώσεις και θα πρέπει να περάσει σε όλα τα καθεστώτα που αναφέρονται στις ευρωπαϊκές περιφέρειες και αυτό απαιτεί χρόνο για την θέσπιση όλων των εργαλείων, όλων των μέσων, ούτω ώστε τα προγράμματα αυτά ε, να μπορούν ε, να εφαρμοστούν όσο το δυνατόν καλύτερα. Λοιπόν, δεν είναι υπερβολικό το αίτημα αυτό για την παροχή λεπτομεριών. Το έχει και επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδιαφέρεται. Θα διαβιβάσω στον ΖΟΑΟ τα αιτήματα των συναδέλφων εδώ για συμπληρωματικά στοιχεία. Θα πρέπει βεβαίως να δούμε ότι δεν πρόκειται για απαγόρευση της αλίας εντός αυτής της ζώνης αλλά απλώ να απαγορεύσει, να απαγορευθούν ε, τα πλοία, τα γρηγρή, ε, που είναι μια σημαντική διαφορά. Αυτή η ζώνη υπάρχει ήδη, η ζώνη προστατευόμενη, υπάρχει ήδη ε, ένα τέτοιο καθεστώς για τις υπερπεριφερειακές ζώνες. Αυτό δεν ξέρω αν οι διευκρινήσεις αυτές είναι σημαντικές σχετικά με το μέγεθος του θαλασσίου πάρκου. Καλύπτει το σύνολο της ζώνης. Η διάσταση αυτή αντιστοιχεί στην οικονομική αποκλειστική ζώνη της Μαγιότ. Μάλιστα, ευχαριστούμε. Κάποια άλλη ερώτηση? Όχι. Είναι αλήθεια ότι είναι κρίμα που δεν είναι εδώ εμπειρογνώμονας. Πάντως, σε ευχαριστώ όλους όσους παρευρίσκεστε. Αλλά θέλω να σας πω ότι το να έρχεστε στην Επιτροπή εδώ του Κοινοβουλίου είναι μία μέρα το μήνα. Έτσι λοιπόν, αν μπορείτε να το προγραμματίσετε κάπως νωρίτερα, θα αποφεύγουμε τέτοιες καταστάσεις. Πάντως τα λέω αυτά στον κύριο Τιπέρη για να τα διαβιβάσει. Να περάσουμε τώρα. Συγγνώμη, προθεσμία κατάθεση τροπολογιών στις 6 Νοεμβρίου το μεσημέρι, 12 το μεσημέρι. Περνάμε στο σημείο 10. Πρωτόκολλο Ευρωπαϊκή Ένωση Μαρόκου για τον καθορισμό ελευτικών δυνατήτων και χρηματική αντιπαροχή που προβλέπουν τη Συμφωνία Ελευτική Σύμπραξη που ισχύει μεταξύ των δύο μερών. Όλοι ξέρετε ότι στι 3 Οκτωβρίου η Επιτροπή και η συγκεντριά μας, η κυρία Φράγκα, έκαναν μια ανταλλαγή απόψεων και σήμερα η κυρία Φράγκα θα μας παρουσιάσει το σχέδιο έκθεσης. Γνωρίζετε πως είχαμε ζητήσει γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας ε, στις 8 του μήνα για θέματα που είχαν τεθεί από την κυρία Λοβίν. Σήμερα εγώ νομίζω ότι ήδη έχει διανεμηθεί η έκθεση της νομικής υπηρεσίας και επομένως ε, έχουν διερευνηθεί όλα τα θέματα τα σχετικά, αλλά σήμερα... Τώρα, τώρα θα πρέπει να το έχετε λογικά. Μοιράζεται τώρα. Μόλις μου το παρέδωσαν εμένα γι' αυτό, σίγουρα και εσείς θα πρέπει να το έχετε. Κυρία Λοβίν. Uh, Ευχαριστώ. Ναι, είναι αλήθεια ότι μοιράστηκε με ε, email ε, πέντε λεπτά μετά την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης ε, και είναι δέκα σελίδες. Ελπίζω λοιπόν να μην θεωρήσουμε ότι έχει ολοκληρωθεί το θέμα αυτό. Θα θέλαμε όμως μια παρουσίαση της νομικής υπηρεσίας και να έχουμε τη δυνατότητα να θέσουμε ερωτήσεις και να στήσουμε διευκρινήσεις. Ευχαριστώ. Εγώ δεν είπα ότι θα το κλείναμε το ζήτημα, απλώς ε, είπα ότι στις 8 Οκτωβρίου είχε ζητηθεί η έκθεση, ότι παραδόθηκε σήμερα και όταν ε, μου το έστειλαν εμένα αμέσω ε, το στείλαμε σε εσείς και όχι μόνο με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αλλά και σε χαρτί θα σας δοθεί εδώ σήμερα. Έτσι λοιπόν, όπως κάνουμε πάντα στις συζητήσεις για οποιοδήποτε θέμα, Φυσικά κατά τη διάρκεια της συζήτησης μπορούν να τεθούν οι ερωτήσεις που θέλετε και στην νομική υπηρεσία αλλά και στην Κομισιόν. Η Προεδρία ποτέ δεν έχει θέσει εμπόδια. Χωρίς χρονοτριβή, η κυρία Φράγκα. Θα προσπαθήσω να μην επαναληφθώ σε σχέση με την τελευταία παρουσίαση που έκανα. Όμως ε, θα επανέλθω σε κάποια από τα σημεία γιατί νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά. Όπως θα θυμάστε και θα επικεντρωθώ και στην έκθεση Χάτλιν που αναλύσαμε τις προάλλες και τις κριτικές που έγιναν στην έκθεση Χάτλιν, Κατόπιν της έκθεσης αυτής έγινε μια πρόταση ψηφίσματος που εγκρίθηκε στην ίδια Ολομέλεια όπου απερίφθη το προηγούμενο πρωτόκολλο και επίσης υπήρχε και μια διαπραγματευτική εντολή του Συμβουλίου. Τόσο η διαπραγματευτική εντολή όπως και η πρόταση ψηφίσματος του Κοινοβουλίου συμπίπτουν σε αρκετά σημεία και κυρίως οι κατευθυντήριες γραμμές διαπραγμάτευσης του Συμβουλίου κάλυψαν αρκετά καλά το θέμα που έπρεπε να διαπραγματευτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακριβώ η εντολή αυτή και η ψηφίσματος αυτό που προσπαθούσαν να κάνουν ήταν να λάβουν υπόψη τις κριτικές που είχαν γίνει στο προηγούμενο πρωτόκολλο. Αν κάποιος δεν θυμάται θα επαναλάβω. Είχαμε το πρόβλημα της οικονομικής αντιπαροχής στη σχέση κόστους-οφέλους που ήταν ένας δείκτης πολύ χαμηλός, ε, τυχή περιβαλλοντική, υπήρχαν αμφιβολίες, σοβαρές αμφιβολίες σε σχέση με τη βιωσιμότητα των πόρων και επίσης ε, την ε, χαμηλή χρήση και υπήρχε και μία άλλη πτυχή που ήταν το πολιτικό ζήτημα για τη Δυτική Σαχάρα. Γιατί, όπως είπε ο κύριος Χάτμουκ, ε, δεν εξέταζε το ζήτημα αυτό καθώς ε, δεν συμπεριλαμβανόταν ε, στους όρους του πρωτοκόλου, όμως ήταν ένα από τα ζητήματα που ανέκυψε κατά τη διάρκεια της συζήτησης εδώ στο Κοινοβούλιο. Η διαπραγματευτική εντολή στο παράρτημα έλεγε τα εξή. Η εντολή, μάλλον, ε, ήταν σημαντική διαπραγματευτική εντολή εγώ πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι είχε μόνο μία αρνητική ψήφο από τη Σουηδία όλες οι άλλες χώρες υπερψήφισαν με τρεις αποχές. Όμως, οι υπόλοιποι υπερψήφισαν, όπως σας είπα, και ζητήθηκε ακριβώς η συμπερίληψη της ε, αλλιευτικής περιοχής νοτίως του παράλληλου 27-40 βορείου δηλαδή τις ζώνες της επικράτειας της Σαχάρας, όπως αποκαλούμε κοινώ. Επίσης, ζητήθηκε ότι προκειμένου να υπάρχει βιώσιμη ανάπτυξη, στόχη της διαπραγμάτευσης θα έπρεπε να είναι η εξή. Η πρόσβαση στους πόρους θα έπρεπε να έχει ως συνέπεια μία επαρκή ανταπόδοση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, χρηματική αντιπεροχή επαρκή και αυτό δεν ίσχυε στο προηγούμενο πρωτόκολλο. Δεύτερο σημείο, να αναλυφθεί δράση για το πλεόνασμα, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και του τοπικού στόλου, όπως και των αλλοδαπών στόλων, πέρα από το δικό μας, το να συμπεριληφθεί στο πρωτόκολλο μία ρήτρα σχετικά με τις συνέπειες σε περίπτωση παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κατόπιν εγγύησης ε, έτσι ώστε το πρωτόκολλο να σέβεται το διεθνές δίκαιο. Και με τις διεθνείς υποχρεώσεις του Μαρόκου στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών. Επίσης ε, ζητούταν σε αυτή την εντολή το Μαρόκο να ενημερώσει για τον κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο της τομεϊκής βοήθειας που προβλεπόταν στο πρωτόκολλο και σε σχέση με τη γεωγραφική κατανομή. Αυτές ήταν οι κατευθυντήριες γραμμές που έλαβε η Κομισιόν και σε πολλές ε, περιπτώσεις εκτός από τα θέματα των υδάτων συμπίπτει με τα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όμως ε, θα αναλύσω τα κυρία σημεία για να δούμε αν ε, έχουν γίνει σεβαστά τα αιτήματα Συμβουλίου και Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά την αποδοτικότητα της συμφωνίας να πω ότι η Κομισιόν έθεσε τη χρηματική αντιπαροχή ε, σύμφωνα με τις ελευτικές δυνατότητες που προσφέρεται. Υπάρχει μείωση 16% στο κόστος που έχει το πρωτόκολλο αυτό σε σχέση με τον κοινοτικό προϋπολογισμό, περνώντας από 36,1 εκατομμύρια ευρώ στα 30 εκατομμύρια ευρώ μειώνεται ο ρυθμός των σκαφών από 137 έχουμε 126 αλλά αυξάνονται οι λευτικές δυνατότητες κατά 33% κυρίως για την κατηγορία 6 που είναι τα πελαγικά είδη, όπου από 60.000 αναβαίνουμε στις 80.000 τόνους. Επίσης υπάρχει αύξηση 5 άδειε στην κατηγορία 2, που είναι ερασιτεχνική αλληλεία. Διορθώνονται τα τεχνικά μέτρα που καθεστούσαν αδύνατο και αυτό ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα που είχαμε στο προηγούμενο πρωτόκολλο. Καθεστούσαν αδύνατο ή δυσκόλευαν τη χρήση ορισμένων κατηγοριών ελίας όπως την κατηγορία 4, κάτι που θα έπρεπε να βελτιώσει τη χρήση αυτού του πρωτοκόλλου χωρίς να θέσει σε κίνδυνο την ε, δεσιμότητα των σκαφών. Κατηγορία 4, παραδείγματο χάρη, προηγούμενος περιορισμός που υπήρχε 270 ε, ήταν ε, ένας από τους λόγους υποεκμετάλλευσης και έτσι ήταν πιο δύσκολο να αλλιεύσουν τα σκάφη πέρα από το ισοβαθές των 200 μέτρων και ήταν αδύνατο λοιπόν να γίνει αλία σε αυτά τα είδατο. γι' αυτό υπήρχε υποεκμετάλλευση αυτής της κατηγορίας. Τώρα τα όρια προσαρμόζονται στα δίδυ σκαφών που χρησιμοποιούν αυτή την κατηγορία και γίνεται μια διαφοροποίηση μεταξύ των σκαφών που αλλιεύουν πελαγικά είδη και τις τράτες ε, και οι τράτες ε, μειώνονται από 11 σε 5. Επίσης διευρύνεται η ελευτική ζώνη για τις κατηγορίες 1 και 2, ρασιτεχνική αλληλεία και φτάνουμε μέχρι το λιμένα της Μοχαμεντία, γιατί εκεί το λιμάνι έχει καλύτερη υποδομή και η υποχρέωση της ε, αποβίβασης θα μπορεί να γίνει, της εκφόρτωσης θα μπορεί να γίνει με καλύτερο τρόπο, γιατί σε άλλα λιμάνια υπήρχαν μεγαλύτερες δυσκολίες. Έτσι λοιπόν, όπως βλέπετε, λαμβάνονται υπόψη μια σειρά τεχνικών ελλημάτων που υπήρχαν και έχουν διορθωθεί σε αυτό το νέο πρωτόκολλο. Τώρα, η αποδοτικότητα της συμφωνίας, αν ε, χρησιμοποιούνταν όλες ε, οι δυνατότητες, αν χρησιμοποιούνταν σε όλες τις δυνατότητες αλία, τις ληφτικές δυνατότητες, ο λόγος που όπως ξέρετε ήταν ε, στο παρελθόν σε λιγότερο από ένα, σε 0,80 κάτι δεν θυμάμαι, τώρα φτάνει στα 2,5 ευρώ. Επομένως, η σχέση κόστους-οφέλους έχει βελτιωθεί τώρα κατά πολύ σε σχέση με την προηγούμενη συμφωνία. Αυτά σε σχέση με την αποδοτικότητα της συμφωνίας, σε σχέση με την αηφορία των πόρων, τη βιωσιμότητα των πόρων και τα περιβαλλοντικά ζητήματα, έχει διανομηθεί μία ενημέρωση από το Μαρόκο που τη ζητήσαμε εμείς ως Επιτροπή και εγώ ως εισηγήτρια για να υπάρχει καλύτερη διαφάνεια για το πώς έγινε ο υπολογισμός αυτός. Η κατηγορία 1 για το στόκ του βορρά των μικρών πελαγικών. Εκεί υπάρχει παρακολούθηση μέσω επιστημονικών εκστρατιών και η ατζούγια είναι 1,8%, ε, η σαρδέλα 1,6%. Έτσι λοιπόν βλέπουμε πολύ μικρό είναι ο αντίκτυπος της αεραστεχνικής αλίας στους Το κύριο θέμα ε, που έχουμε είναι η κατηγορία 6 με τα πελαγικά, ε, βιομηχανική πελαγική αλία. Εκεί η δυνατότητα εκμετάλλευση είναι σχεδόν 1 εκατομμύριο τόνια από τις οποίες το 61% του δυναμικού που είναι δυνατόν να το εκμεταλλευτούμε χρησιμοποιείται τόσο από τους τοπικούς στόλους όπως και από όλους αλλοδαπούς στόλους. Έτσι λοιπόν για αυτή την ποσότητα από, μέχρι να φτάσουμε στο ένα εκατομμύριο του δυναμικού της εκμετάλλευσης προφανώς ε, μας δείχνει ότι έχουμε ένα μεγάλο περιθώριο και οι 20.000 τόνοι που δόθηκαν εκτός στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι που μπορούμε να το αναλάβουμε. επίση στο πρωτόκολλο τίθεται η βάση για τη δημιουργία επιστημονικής συνεργασίας εντατικοποιημένη μεταξύ των δύο μερών που θα καταλήξει σε μια καλύτερη εγγύηση, μεγαλύτερη εγγύηση για την αηφόρο εφαρμογή της συμφωνίας. Το άρθρο 4 του πρωτοκόλου λέγεται ότι δεσμεύονται μέρη να υλοποιούν τακτικά επιστημονικές συνεδριάσεις για να εξετάζουν τα ζητήματα που τίθενται στη Μικτή Επιτροπή και ο μόνιμος χαρακτήρας αυτών των επιστημονικών συμβουλών είναι η μεγάλη καινοτομία σε αυτό το πρωτόκολλο στο παρελθόν αυτός ο μόνιμος χαρακτήρας παροχής επιστημονικών συμβουλών δεν υπήρχε και επομένως αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Επίσης, προκειμένου να εγγυθούμε την αηφορία, τη βιωσιμότητα των ε, αποθεμάτων, Έχουμε εδώ την υποχρέωση για διαχείριση, έλεγχο και παρακολούθηση της ε, αλίας και θα ήθελα να τονίσω την κατάρτιση ενός παραρτήματος σε αυτό το πρωτόκολλο όπου έχουμε ένα ηλεκτρονικό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών όλων των πληροφοριών και των γράφων που σχετίζονται με την τεχνική διαχείριση του πρωτοκόλλου όπως είναι παραδείγματο χάρη οι κοινοποιήσεις για είσοδο και έξοδο ε, από τη ζώνη που βρίσκονται τα σκάφη με το VMS και τα στοιχεία ε, για τα αλλιεύματα και φυσικά αυτό ήταν ένα αίτημα δικό μας παραδοσιακό και βέβαια το Μαρόκο καθώς ε, έχει αναπτυχθεί και αυτό τεχνολογικά μπορούμε τώρα να ε, το υλοποιήσουμε. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα σύστημα πολύ πιο ακριβές και γρήγορο. Σε ό,τι αφορά τώρα την τομεακή πολιτική, τον άρθρο 6 αποτελεί μια πολιτική καινοτομία και απαντά και στις ανησυχίε αυτού του Κοινοβουλίου όπως ε, και τις εντολής του Συμβουλίου. Η τομεακή πολιτική εντάσσεται στην ε, αλευτική στρατηγική και η καινοτομία εδώ στο άρθρο 6 είναι ότι τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να παρουσιαστούν αρκετά εκ των προτέρων και θα υποβληθούν στην έγκριση της Μικτής Επιτροπής, ένα όργανο που θα πρέπει να αξιολογήσει το είναι κατάσταση αξιολόγηση εκτέλεσης των σχεδίων. Θα πρέπει εκεί να αξιολογούνται τα οικονομικά, κοινωνικά, ε, ε, οικονομικές κοινωνικές συνέπειες και επίσης θα λαμβάνεται υπόψη και η γεωγραφική κατανομή. Αυτή την, ε, αυτό το αίτημα το είχε υποβάλει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και το Συμβούλιο και δεν θα γίνει καμία πληρωμή αν δεν αιτιολογηθεί πλήρως ε, ο προορισμός αυτών των κονδυλίων. Έτσι λοιπόν, ε, εγώ ξέρω ότι κάποιοι βουλευτές είπαν ότι δεν τους αρκούσε αυτό, αλλά εγώ πιστεύω ότι αποτελεί σημαντική πρόοδο σε σχέση με τα αιτήματα που υπήρχαν. Δηλαδή, η αξιολόγηση των σχεδίων ανά διάφορες γεωγραφικές ζώνες ε, και μπορούμε να ξέρουμε τι γίνεται στις διάφορες γεωγραφικές περιοχές στο Μαρόκο και ποιος θα είναι ο οικονομικός και κοινωνικός αντίκτυπος αυτών των έργων. Και αυτό σχετίζεται με ένα θέμα που θα δούμε στη συνέχεια. Αν ε, και θέλω να το πω εκ των προτέρων, ε, νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα που και το Κοινοβούλιο αλλά και το Συμβούλιο το έχουν αξιολογήσει Θέλω να επισημάνω ότι στις μεκτές επιτροπές υπάρχει ένας, να υπάρχει ένας παρατηρητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Άπαξ, γιατί η αλήθεια είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την ευθύνη να κάνει αυτές τις εξελογήσεις μεν, αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να έχει έναν έλεγχο αυτού του ζητήματος δε. Επομένω, εγώ θεωρώ ένας εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή κάποιοι εκπρόσωποι θα έπρεπε να συμμετέχουν σε αυτές τις μεικτές επιτροπές. Και το λέω αυτό. Γιατί εγώ ήμουν εκπρόσωπο αυτού του Κοινοβουλίου σε μεικτέ επιτροπέ και για τι συμφωνίε Μαρόκου Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εδώ και δύο-τρία χρόνια Διακόπησε, διακόπηκε αυτή η διαδικασία και δεν μας επιτρέπουν σε εμά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρευρισκόμαστε σε τέτοιες συνεδριάσεις και νομίζω ότι αυτό είναι ένα παράδειγμα όπου θα έπρεπε να επιμπίνουμε εκ νέου γιατί είναι δικαίωμα αυτού του Κοινοβουλίου. Και εδώ ο έλεγχος θα έπρεπε να γίνεται και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και θα επιστρέψω στο θέμα αυτό αλλά θεωρώ ότι είναι σημαντικό να αναφερθώ σε αυτό το σημείο και στο πλαίσιο τη τομεακή πολιτική, ό,τι αφορά τη ρήτρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ξέρετε ότι αυτή ήταν μία από τι εντελέσει τη Κομισιόν, βρίσκεται στο άρθρο 1 του πρωτοκόλου. Και αν ε, σημειωθεί ότι υπάρχει παραβίαση της ρήτρας αυτού, προβλέπεται στο άρθρο 8 η αναστολή της συμφωνίας ε, και της ε, καταβολής της αντίστοιχης χρηματικής αντιπεροχής. Όπως ε, ξέρετε, γίνεται ρητή αναφορά στο άρθρο 2 της Συμφωνίας Σύνδεσης. Ε, γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στο σεβασμό των δημοκρατικών αρχών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και να πω ότι τις ε, προάλλες εξήγησα λεπτομερώς τα άλλα θέματα. Θα περάσω λοιπόν τώρα στο πολιτικό ζήτημα γιατί τις προάλλες δεν ήθελα να παρέμβω, αλλά τώρα θέλω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις αφού διάβασα τις εκθέσεις. Διάβασα και την έκθεση της νομικής υπηρεσίας. Λοιπόν, πολιτικές πτυχές επίσης υπάρχουν στην εντολή του Συμβουλίου. Και ασχολήθηκα εγώ λοιπόν με το θέμα αυτό. Στις κατευθυντήρε γραμμές γίνεται λόγος για το να γίνουν σεβαστέ οι υποχρεώσει από το βασίλειο του Μπαρόκου υποχρεώσεις που έχει αναλάβει έναντι των Ηνωμένων Εθνών. Αυτή ακριβώς είναι η εντολή και πρέπει να ξέρουμε ότι έτσι είναι. ότι το Μαρόκο πρέπει να σεβαστεί αυτές τις υποχρεώσεις. Εγώ θα ήθελα λοιπόν να πω εδώ το εξής. Σύμφωνα με την νομική υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών, και αναφέρομαι στην έκθεση Κόρεν, δεν είναι αντίθετο. Η έκθεση Κόρεν ακριβώς αναφέρεται σε κάποιες ε, πετρελαϊκές εκχωρήσεις σε ύδατα της Δυτικής χάρας ε, στο 2001 που έγιναν από το βασίλειο του Μαρόκου και φυσικά είναι σημαντικό αυτό το θέμα γιατί μιλάμε για ύδατα της Δυτικής Σαχάρας. Έτσι λοιπόν δεν είναι αντίθετο και εγώ λέω ότι εδώ συμφωνεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν είναι αντίθετη εκμετάλλευση πόρων ενός εδάφου με αυτόν, ε, αν γίνεται πάντοτε ε, προς όφελος του πληθυσμού αυτής της επικράτειας. Έτσι λοιπόν ε, και το 2009, η νομική υπηρεσία του 2009, είπε ότι η οθέτηση μιας ελευτική συμφωνίας δεν είναι αντίθετη με το διεθνές δίκαιο και ότι ακριβώς κατά την εκτέλεσή της Δηλαδή, περσέ δεν είναι αντίθετη, αλλά εκτέλεση, η εφαρμογή αυτής της συμφωνίας είναι εκεί όπου μπορούμε να δούμε αν γίνεται σεβαστή όχι νομιμότητα. Δηλαδή, περσέ δεν είναι παράνομη. Αλλά αν στην εφαρμογή της συμφωνίας δεν ε, γίνονται σεβαστές ορισμένες διεθνείς υποχρεώσεις, τότε μπορούμε να κάνουμε τη σχετική αξιολόγηση για το αν είναι νόμιμη ή όχι συμφωνία και θα πρέπει η αξιολόγηση να γίνει στο πλαίσιο της μεικτής Επιτροπής και αν δεν υπάρχει τήρηση των υποχρεώσεων μπορεί να υπάρξει αναστολή της εφαρμογής του πρωτοκόλλου, κάτι που προβλέπεται και στην αναστολή της καταβολής της χρηματικής αντιπαροχής. Έτσι λοιπόν εγώ επιστρέφω στο πόσο σημαντικό είναι το Κοινοβούλιο να έχει και έναν εκπρόσωπο ως παρατηρητή αυτές τις μεικτές επιτροπές για να μπορεί να κάνει έναν έλεγχο να μπορεί να γίνεται και ένας έλεγχος από την πλευρά του Κοινοβουλίου εξάρτητα με το τι κάνει η Κομισιόν για να μπορέσουμε να δούμε αν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της συμφωνίας γίνεται ή όχι σεβαστός ο νόμος, αλλά απριόρι δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι νόμιμη αυτή η συμφωνία. Είναι αλλα πριορι θέμα του πώς εφαρμόζεται αυτή η συμφωνια ειναι το θεμα το πως εφαρμοζεται αυτη η συμφωνια για να οδηγηθούμε στο πορισμά μας. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις που θέλω να κάνω για το θέμα αυτό και κατά τα λοιπά, Πρόεδρε, είμαι στη διάθεσή σας. Έχουμε μοιράσει τα σχετικά έγγραφα, αυτό που μας έστειλε το Μαρόκο και η νομική γνωμοδότηση, πρέπει να τα αξιολογήσετε. Εγώ δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω. Μάλιστα, ευχαριστούμε κυρία Φράγκα. Να δώσω καταρχήν το λόγο στην Κομισιόν και κατόπιν στους υπόλοιπους βουλευτές. Κύριε Δε Yes, uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ την κυρία Φράγκα για την εξαίρετη περιγραφή των όσων διαπραγματευόμαστε. Συμφωνώ πλήρως ότι η εντολή που μας δόθηκε από το Συμβούλιο και οι συστάσεις του Κοινοβουλίου σας ε, συνέκλειναν. Οπότε είχαμε τον κατάλληλο προσανατολισμό, η εντολή ήταν σαφής και βεβαίως ακολουθήσαμε επιμελώς ε, τις συστάσεις και την εντολή. Συμφωνώ με την κυρία Φράγκα ότι αυτό που έχουμε ενώπιόν μας είναι ένα πρωτόκολλο το οποίο βελτιώθηκε πολύ ε, σε σχέση ε, με το κόστος όφελος και η δομή, οι ε, συνεισφορές από το ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για υποστήριξη και από το στόλο μας είναι τέτοιες ώστε τα κίνητρα για τον στόλο να αδειοδοτηθεί ε, και να χρησιμοποιήσει τις άδειες είναι ένα κίνητρο σημαντικό, είναι διαρθρωτική βελτίωση ε, του πρωτοκόλου σχετικά με τις τεχνικές συνθήκες. Πρέπει να πω, αφού διαπραγματεύτηκα με τους Μαροκινούς ότι η προθυμία τους να εξασφαλίσουν οι τεχνικοί όροι να είναι καλοί, να είναι ικανοποιητικοί ούτως ώστε να μην υπάρξουν εμπόδια τεχνικά για την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας. Είναι πολύ καλή συνεργασία. Όσον αφορά επίσης την συνεργασία σχετικά με την επιστημονική ανάλυση, την βιωσιμότητα, ε, έπρεπε εμείς να βεβαιωθούμε ότι όλα αυτά ε, είχαν ικανοποιηθεί και να μην υπάρχουν, έχουμε μη βιωσιμότητα που να παρεμποδίζει την εφαρμογή του πρωτοκόλου και επίσης οι συζητήσεις μεταξύ των επιστημόνων μας και των επιστημόνων τους ήταν πάρα πολύ ικανοποιητικές. Δεν υπάρχει πρόβλημα ε, σχετικά με την βιώσιμη αλία. Έχουμε βεβαίως τεχνικά θέματα ε, τα εργαλεία για τον έλεγχο με ε, συνδυασμό PMS και ERS, ούτως ώστε να ξέρουμε ακριβώς ηλεκτρονικά με τι έχουμε να κάνουμε. Έχουμε ένα πολύ καλό εργαλείο για να βεβαιωθούμε ότι οποιοδήποτε πρόβλημα βιωσιμότητας ε, και αηφορίας θα μπορεί να ανοιχνευτεί πάρα πολύ γρήγορα. Έχουμε λοιπόν ένα πρωτόκολλο το οποίο έχει βελτιωθεί σημαντικά. Το ίδιο σχετικά με τα γεωγραφικά, όπως είπε η κυρία Φράγκα, έχουμε επίση εδώ μία δομή που μας βεβαιώνει ότι θα υπάρξουν αυτές οι αναφορές, η λογοδοσία και θα μπορούμε να συζητούμε τις εκθέσεις και τις αναφορές αυτές. Έχουμε ένα μηχανισμό ο οποίος έχει μεγάλη σημασία και ο οποίος μπορεί επίσης να μας δείξει ότι ότι το θέμα της διεθνούς νομιμότητας δεν θέτει κανένα πρόβλημα. Αυτό το πρωτόκολλο, αυτό καθεαυτό, δεν παρουσιάζει προβλήματα ως προς τη νομική, τη διεθνή νομιμότητα και πρέπει να βεβαιωθούμε ότι η καλή εκτέλεση θα το επιβεβαιώσει αυτό. Θα επιβεβαιώσει λοιπόν, για τους πληθυσμούς και ότι θα έχουμε τα μέσα για το σκοπό αυτό. Θα έλεγα κλείνοντας ότι ένα, μια άποψη ιδιαίτερη αυτού του πρωτοκόλου είναι ότι δεν θέλαμε προσωρινή εφαρμογή, δεν θέλαν και εκείνοι, διότι θέλουν ε, σαφήνεια, θέλουμε σαφήνεια ως προς την ε, προθυμία της Ένωσης να έχει αυτό το πρωτόκολλο που να υποστηρίζεται προτού αρχίσουν οι εργασίες και οι δραστηριότητες. Έπρεπε λοιπόν να βεβαιωθούμε ότι έχουμε το, όλη την, τα μέσα για την εφαρμογή του πρωτοκόλου σχετικά με την ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εκεί νομίζω ότι αυτό που ζητήθηκε για να υπάρχει μια τέτοια διάταξη που να σχετίζεται με τις συνέπειες ε, ως προς προβλήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό αναφέρεται σαφώς ε, στο πρωτόκολλο και υπάρχει, ε, υπάρχει επίσης πρόβλεψη για νομικά μέτρα και βεβαιωθήκαμε με τους εταίρους μας για να δούμε ότι τα όσα εμείς ζητήσαμε και ζήτησε τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς την δυνατότητα αναστολής διακοπής σε περίπτωση προβλημάτων στον τομέα αυτό. Να υπάρχει λοιπόν η πρόβλεψη. Χαίρομαι λοιπόν για τα σχόλια τα οποία έγιναν και είμαι στη διάθεσή σας για περαιτέρω σχόλια. Ευχαριστώ κυρία Λοβίν. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για την έκθεσή της, η οποία είναι πολύ πλήρης. Θα ήθελα να αναφέρω ότι στη σελίδα 7, όσον αφορά την ομιμότητα της συμφωνίας, νομίζω ότι υπάρχει μια ε, λανθασμένη παρατήρηση, διότι λέει ότι η νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου έχει επιβεβαιώσει την ομιμότητα αυτών των συμφωνιών. Και αν ε, κοιτάξουμε την ε, γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου του 2009 είναι απολύτω σαφές ότι η νομική υπηρεσία κατέληξε ότι το πρωτόκολλο θα πρέπει να ανασταλεί. Επειδή δεν υπήρχε καμία απόδειξη, απολύτως, ότι συνάδει με το διεθνές δίκαιο. που ζητάει οποιαδήποτε εκμετάλλευση φυσικών πόρων που ανήκουν σε μία αυτόνομο λαό να ωφελεί τον λαό αυτόν και να χρησιμοποιείται ανάλογα με τις επιθυμίες αυτού του λαού. Αυτό ποτέ, ποτέ δεν έχει θεσπιστεί. Η κυρία Φράγα γνωρίζει καλύτερα από μένα. Δεν διαπιστώθηκε μάλλον αυτό. Η κυρία Φράγα γνωρίζει ότι το 2010 η Επιτροπή μας προσπάθησε να οργανώσει αποστολή στο Μαρόκο και να επισκεφτεί και τη Δυτική Σαχάρα, να συναντήσει τους ανθρώπους για να διαπιστώσουμε με τα μάτια μας εάν η Συμφωνία Αλίας με το Μαρόκο ωφελεί τους ανθρώπους της Δυτικής Σαχάρας. Δεν μας επέτρεψαν όμως να έρθουμε. Εκτιμώ την πρόταση της κυρίας Φράγα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να μπορέσει να να μπορεί να συμμετέχει στις ε, κοινέ επιστημονικές συνεδριάσεις. Ε, νομίζω ότι πραγματικά ε, είναι περίεργο το ότι δεν μπορούμε να συμμετέχουμε, αλλά αμφιβάλλω αν θα... αν θα λαμβάνουμε περισσότερες επιστημονικές πληροφορίες στις συναντήσεις αυτές από ό,τι έχει καταφέρει να λάβει η Κομισιόν. Ξέρω ότι επί χρόνια προσπαθούσαμε στην Επιτροπή μας να βρούμε αποδείξεις από το Μαρόκο σχετικά με την κατανομή των οφελών ε, των αλληλευτικών συμφωνιών, με τον τρόπο που το παρουσιάζει το Μαρόκο, σε γεωγραφικούς όρους δηλαδή, με γεωγραφικούς όρους. Ε, και θυμάμαι ότι ήταν εδώ η Επίτροπος Μαρία Δαμανάκη, η οποία επανειλημμένα εξήγησε στην Επιτροπή μας ότι η Επιτροπή δεν έχει λάβει πληροφορίες. Και τελικά μετά από πάνω από ένα χρόνο έλαβε το Κοινοβούλιο πληροφορίες εμπιστευτικές. Μπορούσαμε λοιπόν να πάμε στη γραμματεία να υπογράψουμε και να δούμε τις πληροφορίες που ε, ήρθαν από το Μαρόκο. Οι πληροφορίες του Μαρόκο ήταν ε, μία παρουσίαση PowerPoint, η οποία δεν εξηγούσε πολύ αναλυτικά τη νέα στρατηγική αλίας του Μαρόκου και κατόπιν εξηγούσε κάπως τη γεωγραφική κατανομή των επενδύσεων. Δεν αναφερόταν όμως συγκεκριμένα στο θέμα της Δυτικής Σαχάρας και το πώς η συμφωνία αυτή θα ωφελούσε τους ανθρώπους της Δυτικής Σαχάρας. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια νομική γνωμοδότηση του Χαν Κορέλ των Ηνωμένων Εθνών που τονίζει ότι δεν είναι, δεν είναι δεν αρκεί ακόμα και αν διαπιστώσουμε ότι η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων ε, ε, ωφελεί έναν μη αυτόνομα λαό, ε, διότι θα πρέπει να τους ωφελεί σύμφωνα με τις επιθυμίες τους και αυτό δεν έχει διαπιστωθεί καθόλου. Αντιθέτως, στην τελευταία ε, συνάντηση με την Επιτροπή. Ε, στην ε, απολύτως σαφή και αυτή απάντηση, εάν έχετε συναντηθεί με εκπροσώπους της Δυτικής Σαχάρας, μας είπαν ότι ναι, έχουμε συναντηθεί και... Ξέρουμε τι λένε, διότι σήμερα έχω λάβει email, ηλεκτρονικό μήνυμα από έναν εκπρόσωπο τουλάχιστον Μπορεί κάποιος να αμφισβητήσει αν το Πολυσάριο ε, εκπροσωπεί όλους ε, τους ανθρώπους της Δυτικής Σαχάρας, αλλά ε, εκπροσωπεί σημαντική πλειοψηφία του λαού αυτού. Ο Μοχάμετ Απτελασής, λοιπόν, γράφει προς όλα τα μέλη της Επιτροπής μας και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ως η υπερεθνική ένωση που βασίζεται στην ελευθερία, την τα ανθρώπινα δικαιώματα κλπ. δεν θα πρέπει να συμμετέχει στην κλοπή ε, που πραγματοποιείται. Ε, είναι λοιπόν απολύτως σαφές ότι δεν έχει γίνει διαβούλευση με τους ανθρώπους αυτούς και δεν έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους ε, για την εκμετάλλευση αυτή. Ας πάμε λοιπόν πίσω στο τι είπε το Κοινοβούλιο στην... στο περίφημο ψήφισμα που υιοθετήθηκε Όταν, είπαμε, όταν απορρίψαμε την έκθεση Χάγκλοντ, όταν είπαμε ε, όχι στην ε, Συμφωνία Λίας. Το έλεγξα σήμερα. κοιτάξτε κοιτάξετε την ε, παράγραφο 3, λέει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διασφαλίζει ότι τα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν πρόσβαση μόνο σε κάποια αποθέματα και τονίζει ότι θα πρέπει να γίνει αξιολόγηση, αυστηρή αξιολόγηση όλων των αποθεμάτων. Και παρότι έχουμε λάβει τόσες νέες πληροφορίες ε, σήμερα από το Μαρόκο σχετικά με τα αλληλευτικά αποθέματα, θα πρέπει να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί δεν εξέτασε την παράγραφο 10, όπου ζητάμε από την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο γραπτή αναλυτική έκθεση που να δείχνει το βαθμό που έχουν ληφθεί υπόψη οι επιθυμίες του Κοινοβουλίου για το μελλοντικό πρωτόκολλο. Ζητάμε λοιπόν γραπτή έκθεση και νομίζω ότι μια τέτοια έκθεση θα είναι πολύ χρήσιμη όταν μιλάμε για τόσο πολύπλοκα πράγματα όσο είναι η αξιολόγηση των αποθεμάτων κλπ. Δεν έχουμε λάβει τα ε, στοιχεία αυτά, μόνο κάποιε φήμε έχουμε ακούσει. Τώρα λοιπόν έχουμε τι πληροφορίες αυτέ από το Μαρόκο. Εγώ θα εκτιμούσα πάρα πολύ να λάβω μια ανάλυση σχετικά με την κατάσταση των αποθεμάτων, διότι φαίνεται να είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό για πολλού ευρωβουλευτέ. Στην παράγραφο 8 Ζητάμε από την Επιτροπή να εισάγει στην ε, Αλλιευτική Συμφωνία ε, μία ρήτρα συμμόρφωσης ε, με τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως αναφέρεται στο ψήφισμα του 2010 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και κοινωνικοπεριβαλλοντικά πρότυπα σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες. Έψαξα λοιπόν να βρω το ψήφισμα αυτό και στο ψήφισμα αυτό λέει ότι στηρίζει την πρακτική να συμπεριλαμβάνονται δεσμευτικές ε, ρήτρε ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις εμπορικές συμφωνίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα ήθελα και πάλι να τονίσω ότι μιλάμε για νομικά δεσμευτικές ρήτρες, διότι αυτό που βλέπουμε στο πρωτόκολλο αυτό είναι μια πολύ χαλαρή αναφορά στις, ε, ε, στην Συμφωνία Σύνδεσης ε, και διαφωνώ απολύτως με όποιον λέει ότι αυτή είναι ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν είναι. Η ρήτρα αναστολής είναι τελείως διαφορετική και δεν συνδέεται με το θέμα αυτό. Και αν κοιτάξουμε την Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Μαρόκου, δεν λέει πουθενά ότι είναι νομικά δεσμευτικό το να ακολουθεί κανεί ε, τον ε, χάρτη των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Λέει ότι είναι εμπνευσμένο. Εμπνευσμένο. Αυτό είναι το, το, ρήμα που χρησιμοποιείται. Και αυτή είναι πολύ σημαντική διαφορά. Όλα λοιπόν τα μέλη της Επιτροπής μας, ε, ε κάθομαστε εδώ, ακούμε την Επιτροπή, επί μήνες να μα εξηγεί πώ προχωράνε οι διαπραγματεύσει Ευρωπαϊκή Ένωση Μαρόκου. Και ακούσαμε ότι ένα από τα σημαντικά εμπόδια ήταν η συμπερίληψη μια ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το έχουμε ακούσει αυτό από την Επίτροπο. Το, αυτό ακούμε συνέχεια. Το ποσό χρημάτων και η συμπερίληψη ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και γιατί είναι τόσο ε, ε, ε, ευαίσθητο το θέμα αυτό για το Μαρόκο. Τη στιγμή που αυτό αποτελεί μέρος οποιασδήποτε ε, συμφωνίας αλλίας που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να το αναρωτηθούμε αυτό. Και επίσης αναρωτιέμαι γιατί το Μαρόκο δεν καλωσόρισε την ε, Επιτροπή μας ε, στην, ε, στο Μαρόκο, γιατί δεν θεώρησε ευπρόσδεκτη την Επιτροπή μας στο Μαρόκο για να δούμε με τα μάτια μας τι ακριβώς συμβαίνει. Και γιατί δεν επιτράπει στα μέλη του Κοινοβουλίου να επισκοφτούμε τις κατεχόμενες περιοχές για να δούμε με τα μάτια μας τι συμβαίνει εκεί. Παρότι σαφώς το αναφέραμε αυτό, ενημερώσαμε τον πρέσβη σχετικά με τις προθέσεις μας. Θελήσαμε να επισκεφτούμε τις ε, μαροκινές αρχές ε, και δεν ε, μας το επέτρεψαν. Εγώ είμαι περήφανη για το κοινοβούλιο μας, διότι είναι ένα μέρος όπου επικρατεί διαφάνεια. Μπορεί κανείς να παρακολουθήσει στο ίντερνετ, σε απευθεία μετάδοση την συνεδρίαση αυτή. Έχουμε πολλούς εκπροσώπους από το Μαρόκο αυτή τη στιγμή στην αίθουσα. Ποιο θα παρακολουθήσει την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Δυτική Σαχάρα, αν δεν επιτρέπεται σε κανέναν να πάει εκεί. Η Κομισιόν παρακολουθεί τα θέματα αυτά. Θα παρακολουθήσετε την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Δυτική Σαχάρα. Η εκπρόσωποι τη ε, Γενική Διεύθυνση ε, για τη Θάλασσα, Μάρε, λέει ότι δεν είμαστε εμεί εμπειρογνώμονε για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ποιο θα το κάνει αυτό λοιπόν. Και τι είδου αξιολόγηση θα γίνει. Η τελευταία έκθεση του εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών ε, για τα βασανιστήρια και ε, ε, ε, άλλων ειδών κακής απαξιωτικής μεταχείρισης κλπ. Ποιο ακούμε εμεί, πώ θα παρακολουθήσουμε την κατάσταση αυτή. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ασαφή τα πράγματα και νομίζω. ότι η άποψη των τη ε, της νομικής υπηρεσίας και έχουμε λάβει τώρα την νέα γνωμοδότηση είναι ότι αν δεν μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι η εφαρμογή γίνεται ανάλογα με τις επιθυμίες και προς όφελος του τοπικού πληθυσμού δεν είναι νόμιμη. Με αυτά θα κλείσω διότι θα ήθελα η Επιτροπή μας να έχει την ε, ευκαιρία και το χρόνο να ακούσουμε παρουσίαση της ε, νέας, νομικής, ε, της νέας νομοδότησης νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου σχετικά με το αν το Μαρόκο έχει το δικαίωμα να, να πουλάει τους αλληλευτικούς πόρους της Δυτικής Σαχάρας και πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε το χρόνο για να σκεφτούμε τη συμφωνία αυτή, να μην βιαστούμε να κάνουμε κάτι, να μην ψηφίσουμε προτού να ε, έχουμε παρουσίαση της ε, γνωμοδότησης ε, στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρωμέδα. Ευχαριστώ. Εγώ δεν θα μακρηγορήσω γιατί συμφωνώ με όλα εσύ που μόλις συνάδελφος. Καταρχήν θέλω να κάνω μια ερώτηση. Δεν ε, θυμάμαι ποτέ να έχει τεθεί ερώτηση εδώ σε αυτό τον ε, οίκο από ποιο κόμμα προέρχεται ένας ε, συνάδελφος από το Μαρόκο για να μπορεί να παρευρεθεί σε μια συνεδρίαση. Και το λέω αυτό η για να μπει Το λέω γιατί Κάθε φορά εμείς που πάμε στο Μαρόκο αυτό συμβαίνει από την άλλη πλευρά. Ε, δηλαδή όταν ε, περνά ένας Μαροκινός στα σύνορα, δεν τον ρωτάμε για τις πολιτικές υπευθύσεις αλλά και σε μένα και στη συνάδελφο στην κυρία ε, Λοβίν, τέθηκε αυτό το ερώτημα και εγώ νομίζω ότι είναι πολιτικά ευαίσθητο και μας εκπλήσει βεβαίως. Λοιπόν, σύμφωνα με όσα είπε η κυρία Λοβίν και ξέρω ότι σήμερα έχουμε πολλούς συναδέλφους από το Μαρόκο που σίγουρα θα αναρωτηθούν γιατί κάποιοι ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ να είναι ανοιχτό αυτό το θέμα και να είναι δημόσιο, γιατί δεν μπορούμε πάντοτε να το κάνουμε αυτό όταν μιλάμε για θέματα που αυτούς τους ενδιαφέρουν. Ένα δεύτερο θέμα που θέλω να τονίσω και μου φαίνεται σημαντικό είναι το αξίζει Έχουμε ένα ντεζαβού εδώ Δηλαδή έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση χιλιάδες φορές και υπάρχει ένα θέμα που συνεχίζει ανεπίλητο. Υπάρχει και ένα σημείο που το έθεσε και η κυρία Φράγκα, δηλαδή τίθεται ότι δεν είναι παράνομο το κείμενο και το είπε και η Κομισιόν. Από την άλλη όμως υπάρχει μια αντίφαση μεταξύ του τι λέγεται και του τι συμβαίνει όταν ακριβώς ε, τίθεται το θέμα ότι η νομιμότητα βασίζεται στο να ευνοεί η πολιτική που εφαρμόζεται τον πληθυσμό της Δυτικής Σαχάρας αφενός και από την άλλη ε, βλέπουμε ρητά ότι ένα από τα μέρη που άμεσα συμμετέχουν στη διαδικασία και μας δηλώνει, το Πολυσάριο λοιπόν μας δηλώνει ότι ποτέ δεν έχει ζητηθεί η δική του γνώμη και μάλιστα τα όσα γίνονται είναι και κατά των συμφερόντων του. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένα πρόβλημα ουσιαστικό εδώ και εγώ θα ήθελα τουλάχιστον να είναι ξεκάθαρο το εξή. Οι κυβερνήσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κομισιόν ουσιαστικά παίζουν το παιχνίδι της κυβέρνησης του Μαρόκου χρησιμοποιώντας την αλία. Πάντοτε εδώ μας λένε ότι σε αυτήν την επιτροπή συζητάμε θέματα αλίας και όχι για να κάνουμε πολιτική, κάτι που είναι παράδοξο, γιατί στο Κοινοβούλιο γίνεται πολιτική σε όλες τις επιτροπές. Όμως, αν ειδικά σε κάποιο κείμενο γίνεται πολιτική, είναι ακριβώς σε αυτό εδώ, γιατί αυτό που θέλει το Μαρόκο είναι πολύ απλό ως Ευρωπαϊκή Ένωση και ως Κοινοβούλιο να επικυρώσουμε την πολιτική που ακολουθεί με τη Δική Σαχάρα. Ε, ούτε λιγότερο, ούτε περισσότερο, είτε μας αρέσει είτε όχι. Σε κάποιους δεν αρέσει, αλλά αυτό γίνεται. Και η Κομισιόν και κυρίως κάποιες κυβερνήσεις της Ισπανίας και της Γαλλίας ακριβώς αυτό κάνουν τώρα. Τι ζητάμε ορισμένες ομάδες. Ορισμένες ομάδες ζητάμε κάτι πολύ απλό που μάλιστα ήδη έχει γίνει σε άλλες συμφωνίες, παραδείγματος χάρη μεταξύ Μαρόκου και Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή ρητός να αποκλειστούν τα εγχώρια ύδατα ε, το, της Δυτικής Σαχάρας από το πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας. Και αυτό έχει να κάνει με την πολιτική βούληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εγώ αναρωτιέμαι μετά από τόσα χρόνια που το συζητάμε, γιατί δεν έχει γίνει. Είναι πολύ απλό. Είναι πολύ απλό. Αν δεν συμφωνήσουμε για την νομική διάσταση της εκμετάλλευσης ε, των ε, εγχώριων υδάτων της Δυτικής Σαχάρας, η λύση έγκυται και το λέει και η νομική σύσταση του Συμβουλίου, έγκυται στο ότι αν δεν υπάρχει μια φιλική συμφωνία μεταξύ των μερών, να αποκλειστούν ε, από τη συμφωνία τα ύδατα της θετική Σαχάρας. Αυτή είναι η ερώτησή μου λοιπόν και θα ήθελα να μας εξηγήσει και η Κομισιόν γιατί δεν έχει γίνει ακόμη και γιατί σήμερα εξακολουθούμε να μιλάμε αόριστα. Θα ήταν ε, πάρα πολύ εύκολο και θα εξοικονομούσαμε ώρες επί ωρών συζήτησης. Εμένα λένε κάτι και οι άλλοι το αντίθετο και γιατί δεν το κάναμε αυτό για να τελειώνουμε και Τώρα από εδώ και πέρα συζητάμε τι θα κάνουμε με τη διαχείριση μία συμφωνία ε, με εκείνα τα χωρικά ύδατα τη Δυτική Σαχάρας. Αλλά εμείς ε, όσο δεν επιλέγεται αυτή η λύση θα είμαστε αντίθετοι σε αυτή τη συμφωνία γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει και το διεθνές δίκαιο σεβαστό. Ευχαριστώ κύριε Ρωμέβα και κυρία Πατράου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μετά την παρουσίαση της κυρίας Φράγκα, για αυτή την πρόταση συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μαρόκου, δεν υπάρχουν πολλά να προσθέσω. Ήταν ιδιαίτερα πλήρης και λεπτομερής η παρουσίαση. Και Για τα αντεπιχειρήματα εγώ δεν νομίζω ότι χαίρουν ε, και μια λογική βάση. Ο ευρωπαϊκό στόλο έχει ζημιωθεί πάρα πολύ ε, σε σχέση με το τι συνέβη το 2011. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο κλάδος της επίσης έχουν ζημιωθεί, αλλά Επίσης ε, και οι πόροι που διαθέτει το Μαρόκο για συμφωνίες με άλλες χώρες ε, συνεχίζουν να είναι αντικείμενο αλίας και ξέρετε ότι οι συνθήκες είναι πολύ διαφορετικές από αυτές που θα έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα παντού σε ολόκληρο τον κόσμο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τις μεγαλύτερες απαιτήσεις για τη θέσπιση συμφωνιών με τρίτες χώρες. Και ε, ακόμη και αν είναι αυτά τα μοντέλα απαιτητικά, υπάρχουν πολλές δυσκολίες και φυσικά αυτό ζημιώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον κλάδο της Ελίας και δεν φέρει κανένα όφελος, κυρίως και ως προς ε, αυτά που υπερσπιζόμαστε. Και, και αυτό είναι ένα ακόμα παράδειγμα. Τώρα, η συμφωνία που έχουμε τάπητος είναι πάρα πολύ ισορροπημένη. Και σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα των πόρων, τις ελευτικές ικανότητες, τη χρηματική αντιπαροχή. και όλες αυτές τις πτυχές, η συμφωνία αυτή πραγματικά ωφελεί και τα δύο μέρη. Και εμάς Φυσικά εδώ μας ενδιαφέρει κυρίως να αφαιρεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί έχουμε πει ότι εδώ εμείς ε, θέλουμε να υπερασπίσουμε τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν υπάρχει καμία ότι τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα υπερασπιζόμαστε πάρα πολύ καλά με αυτήν την πρώτη συμφωνία που έχουμε ενωπιό μας. Τώρα δεν θέλω να μακρηγορήσω γιατί απλώς ε, θα επαναλάμβανα όσα υπόθηκαν από την συγγήτρια γιατί ήταν ιδιαίτερα εξαντλητική η παρουσίασή τη. Θα ήθελα ωστόσο να υπογραμμίσω δύο πτυχές που πιστεύω ότι δεν υπογραμμίστηκαν αρκετά. Το πρώτο έχει να κάνει με το γεγονός ότι το 2011 εμείς ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίναμε ένα ψήφισμα που είναι η δική μας δέσμευση με το Μαρόκο και η συμφωνία αυτή ε, ουσιαστικά πλήρως ε, ακολουθήθηκε. Αυτή η συμφωνία ήταν μια δέσμευση που εμεί αναλάβαμε για αυτό το θέμα και η συμφωνία που έχουμε ενωπιών μας αυτή τη στιγμή σέβεται σε όλα τα επίπεδα το ψήφισμα που εγκρίναμε εμείς οι ίδιοι. Αυτό δεν μπορούμε να το μελήσουμε. Το δεύτερο που θα ήθελα να υπογραμμίσω έχει να κάνει με τη ρήτρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που επίσης συνάδει με τη Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Μαρόκου. Και από νομική σκοπιά είναι σημαντική αυτή η ρήτρα και μας δίνει επαρκείς εγγύησης και αποτελεί σίγουρα ένα βήμα προς τα μπρος σε σχέση με αυτά που είχαμε το 2011. Και τέλος. Νομίζω ότι πρέπει να τονιστεί και το εξή, ότι μία από τις μεγάλες ανησυχίε της Επιτροπής Ελίας είχε να κάνει με το να εγγυθούμε τη βιωσιμότητα των πόρων και επί της πτυχής αυτής η συμφωνία που έχουμε πει τάπητος είναι παραδειγματική γιατί υπάρχουν όλες οι απαιτήσει επιστημονικής παρακολούθησης ε, ολόκληρης ε, της διαδικασίας και καθόλου τα τέσσερα έτη που θα διαρκέσει η συμφωνία. Και αυτό αποτελεί σημαντικό βήμα προς τα μπρος που δίνεται με αυτή τη συμφωνία και θα μπορούσε να αποτελέσει και παράδειγμα για άλλες συμφωνίες που θα αξιολογήσουμε εμείς εδώ. Σας ευχαριστώ και θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Φράγκα για την εξαιρετική δουλειά της. Ευχαριστώ κύριε Πατράου, επόμενος ομιλητή. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος. Και θα μιλήσω ειδικά εφόσον έχω αυτή τη δυνατότητα. Θα είμαι πολύ σύντομος, διότι επί της αρχής ε, συμφωνώ με αυτά που είπε η Ισαμπέλα Λεβίν θα πρέπει να σκεφτούμε τι ισχύει στο, εθνικό, στο διεθνές δίκαιο και ε, ποιος το ερμηνεύει. Ε, τα Ηνωμένα Έθνη το ερμηνεύουν και έχουμε μια ε, ε, παράνομη κατοχή της Δυτικής Σαχάρας. Αυτό είναι το σημείο εκκίνησης. Δεν μπορούμε να υπογράψουμε συμφωνία με το Μαρόκο εάν δεν αποκλείσουμε το κομμάτι που ανήκει στους ε, ανθρώπους της ε, Δυτικής Σαχάρας. Στην ε, Σουηδία όλα τα κόμματα σύμφωνουν σε αυτό. Και η κυβέρνηση. Είναι λοιπόν ένα θέμα στο οποίο δεν διαφωνεί κανείς. Και πιστεύω ότι και στην Ολομέλεια την ίδια συζήτηση θα έχουμε. Θα έχουμε πλειοψηφία η οποία θα απορρίψει το πρωτόκολλο για του ίδιου λόγου που αυτό έγινε την προηγούμενη φορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Βίλσον. σαν Πρισέδο. Ευχαριστώ. Ήδη έχει επαναληφθεί αυτή η συζήτηση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιοι από τους λόγους που εκφράστηκαν στο παρελθόν δεν έχουν αξία τώρα. Και επίσης ε, ότι δεν είμαστε ικανοί να αξιολογήσουμε τις καινοτομίε που υπάρχουν στο σημερινό πρωτοκολλό. Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι άκουσα πολύ προσεκτικά και είμαι πολύ ευαισθητοποιημένος για τις πολιτικές πτυχές. Εγώ νομίζω ότι το Μαρόκο είναι ένας γείτονα με τον οποίο θέλουμε να έχουμε προνομιακές σχέσεις ε, και να συμβάλλουμε και στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και των δύο μερών. Ε, πριν ε, ένα χρόνο περίπου εγκρίναμε μια συμφωνία για τα γεωργικά προϊόντα και είναι προφανές ότι θα πρέπει σε ένα πνεύμα συνεργασίας θα πρέπει να λυθούν τα πολιτικά ζητήματα με το Μαρόκο που είναι ε, ο πιο σημαντικός γείτονάς μας από την άλλη όχθη της Μεσογείου. Εγώ ήθελα να πω ότι κάποιες από τις ανησυχίες που έχουν τεθεί και στο παρελθόν Νομίζω ότι τώρα απαντήθηκαν πραγματικά. Επιτυχία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ένα από τα σημαντικά θέματα της νέας ελευτικής πολιτικής έχουμε ρητή αναφορά στο άρθρο 1 και υπάρχει και στο άρθρο 8 η αναφορά στην αναστολή της συμφωνίας. Επίσης ε, ε, αυτό έχει να κάνει και με τη συμφωνία σύνδεσης που έχουμε με το Μαρόκο, η οικονομική ανισορροπία. Επίσης υπάρχει μικρότερη ευρωπαϊκή συνεισφορά, ενώ ταυτόχρονα αυξήθηκε η τομεκή στήριξη Υπάρχει μείωση λοιπόν της ευρωπαϊκής συνεισφοράς, υπάρχουν κάποιες ανησυχίες περιβαλλοντικού χαρακτήρα, υπάρχει μείωση του αριθμού των σκαφών, περνάμε, από τα 120, περνάμε στα 127 από τα 136, υπάρχει και τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών. Υπάρχει λοιπόν εδώ μια εξέλιξη, έχουν αντιμετωπιστεί ανησυχίες του Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίου. Υπάρχει όμως και μια πτυχή που θα ήθελα να αναφέρω και έχει να κάνει με τη διεθνή νομιμότητα. Εγώ ως βουλευτής από την Ισπανία θέλω να πω ότι η Ισπανία είναι μια χώρα η οποία πάντοτε ήταν ευαίσθητη σε αυτό το πρόβλημα είναι η χώρα που συνεργάζεται περισσότερο με το λαό της Δικής Σαχάρας ε, και υποδέχεται πολλές, φαμ... Ε, πολλές οικογένειες από την ε, Σαχάρα και τις εντάσεις της ευρωανικές οικογένειες. Επομένως θέλουμε να συνεισφέρουμε στην επίλυση αυτού του προβλήματος. Εγώ νομίζω όμως ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι παράνομο κατά κάποιο τρόπο το πρωτόκολλο. Και είδαμε και το κείμενο που λάβουμε σήμερα, το οποίο λέει ότι δεν υπάρχει καμία ρήτρα που να καθιστά το κείμενο παράνομο διεθνές. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε αυτές τις πολιτικές συμφωνίες σε ένα άλλο πλαίσιο θα πρέπει αυτές οι ανανεώσιμες πηγές να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βελτιωθεί ή για να βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής των ανθρώπων εκεί. Και εμείς αυτό θέλουμε να κάνουμε, ούτε οι Ηνωμένε Πολιτείε, ούτε άλλες χώρες που έχουν αλλιεύσει ποτέ σε αυτές τις περιοχές, το τι θα συμβεί τους είναι τελείως αδιάφορο, όμως υπάρχουν στόλοι που ε, συνεισφέρουν στην ανάπτυξη αυτών των κοινοτήτων και μπορούν να συνεισφέρουν στην ανέβρεση λύσεων που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα καλύτερο κλίμα για το πολιτικό ζήτημα, για την επίλυση του πολιτικού ζητήματος. Εμείς υπερασπίζουμε την αυτοδιάθεση ε, της δυτικής, του λαού της Δυτικής Σαχάρας. Πιστεύουμε ότι αυτό το θέμα πρέπει να επιληθεί στα πλαίσια του ΟΗΕ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεισφέρει για να γίνει πρόοδο στο ζήτημα αυτό και θεωρούμε ότι το σημερινό πρωτόκολλο αποτελεί μια καλή λύση. Αποτελεί ένα ισορροπημένο πρωτόκολλο για το θέμα της Ελίας και σέβεται και τη διεθνή νομιμότητα. Ευχαριστώ κύριε Σάντσες Πρεσέδο, κύριο Καντέκ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ πλήρως με τον συνάδελφο. Είμαστε εδώ για να κάνουμε πολιτική. Γι' αυτό έχουμε εκλεγεί. Και είναι ο λόγος για τον οποίο πιστεύω ότι η συμφωνία αυτή είναι καλή συμφωνία, διότι ακριβώς κάνω πολιτική. Αυτή η συμφωνία θα πρέπει ε, να ωφελεί όλους, όλα τα εδάφη. Βεβαίως τα προβλήματα ανάμεσα στη Δυτική Σαχάρα ε, και το βασίλειο του Μαρόκου υπάρχουν, αλλά όπως λέχθηκε με πάρα πολύ συνεκτικότητα από τον συνάδελφο, έχουμε εδώ ενώπιόν μας μια συμφωνία που είναι καλή συμφωνία και εγώ επιθυμώ να ευχαριστήσω την συνάδελφο Κάρμεν για όλη την εργασία που έκανε σχετικά με το φάκελο αυτό μεταξύ αυτών που υποστήριξαν την προηγούμενη συμφωνία στην εταιρική σχέση με το Μαρόκο και υποστηρίζω αυτή τη νέα συμφωνία. Δεν ξέρω αλλά ελπίζω ότι η πλειονότητα των συναδέλφων, η πλειοψηφία θα υποστηρίξει τη συμφωνία αυτή. Υπάρχουν μερικές πρόοδοι, στη ε, συνεργασία Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, οι κατηγορίες είναι ίδιες, έχουμε αύξηση 33%, ε, προσαρμόστηκαν στην πραγματική χρήση από τους επαγγελματίες ως πρωτατεχνικά μέτρα. Έχουν γίνει δεκτά τα αιτήματα στο πλαίσιο του πρωτοκόλου για τις επιτρεπόμενες ζώνες. Έχουμε επίσης τον αριθμό ε, των ναυτικών ε, στα πλοία που έχει αυξηθεί ε, ανεξάρτητα από την γεωγραφική προέλευση, είτε προέρχονται είτε είναι Σαχράουι είτε προέρχονται από το Μαρόκο. Σχετικά με την ρήτρα σεβασμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αυτή η ρήτρα έχει ενισχυθεί, ήμασταν όλοι υπέρ της ενίσχυσης αυτής, κυρίως η μη, ο μη σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή ε, της εφαρμογής ε, του πρωτοκόλου. Και θα πρέπει το Μαρόκο ε, να δικαιολογεί τις επιλογές του για την χρησιμοποίηση αυτής της ενίσχυσης, της βοήθειας. Νομίζω ότι είναι μια συμφωνία που λαμβάνει υπόψη της. Ε, ε, τα οικονομικά αιτήματα ε, κοινωνικά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γι' αυτό υποστηρίζω πλήρως τη συμφωνία αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Στόρβαλτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Φράγκα για την εργασία της, για την εισήγησή της Είχαμε μακροσκελή συζήτηση για το θέμα αυτό στην ανταλλαγή απόψεων πριν από μερικές εβδομάδες. Γι' αυτό θα αναφερθώ σε συγκεκριμένα σημεία. Δεν μπορώ να ακολουθήσω την σύσταση της ε, Κάρμεν ε, για συνένεση από το Κοινοβούλιο για τους επόμενους λόγους. Έχουμε ε, πάρα πολλές ανησυχίες σχετικά με το περιβάλλον, με τα αποθέματα δεν έχουμε σαφή απόδειξη ότι έχουν βελτιωθεί τα αποθέματα, ενώ θα έπρεπε να έχουμε αυτή την απόδειξη πρωτού προχωρήσουμε με το πρωτόκολλο. Δεύτερον, ε, έχουμε την αξία για το χρήμα ε, που δίδεται. Βεβαίως, ε, τα τέλη που θα πληρώσουν οι εφοπλιστές είναι πολύ μεγαλύτερα, διότι έχουν μεγαλύτερο κέρδος, ποσοστό κέρδος. Δεν ξέρω αν ο φορολογούμενος ε, θα ωφεληθεί. Τρίτον, και αυτό είναι το σημαντικότερο θέμα, δεν ε, σεβόμαστε τη Δυτική Σαχάρα και τα ανθρώπινα ε, δικαιώματα. Όλοι από εσά θα θυμάστε όταν είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής, όταν μίλησε για την κατάσταση της Ένωσης, μίλησε πολύ για τις αξίες, αλλά συνήθως προσκρούμε στο ίδιο πρόβλημα. Ε, μιλάμε τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις Αργίες για τις αξίες και όταν επανερχόμεθα στην πραγματικότητα βλέπουμε ότι ξεχνούμε τις αξίες. Έχουμε άλλα κράτη όπως ε, τα Ηνωμένε Πολιτείες ε, Βεβαίω βλέπουμε τι κάνει στις συμφωνίες με το βασίλειο του Μαρόκου και την ε, Δυτική Σαχάρα. Το ίδιο γίνεται και από άλλες χώρες. Και εμείς ε, θα πρέπει να κάνουμε το ίδιο πράγμα. Παρόλο που το θέμα αυτό δεν αναφέρθηκε ρητά στην έκθεση Χάγκλουντ, το θέμα της Δυτικής Σαχάρας υπάρχει πάντοτε και είναι σημαντικό θέμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να έχει διπλά μέτρα και σταθμά όταν πρόκειται για τα ανθρώπινα δικαιώματα και αυτό πρέπει να ισχύει για την Επιτροπή Ελίας. Μιλούμε, κάνουμε κηρύγματα ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον δυτικό κόσμο με τρόπο που συχνά δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και μια συμφωνία που δεν θα σεβόταν τη Δυτική Σαχάρα θα ερχόταν σε αντίφαση με τα όσα κηρύσουμε. Δεν πρέπει να αποκλείονται λοιπόν τα ύδατα της Δυτικής Σαχάρας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καπουλασάντος. Και εγώ καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Φράγα για το έργο της. Και νομίζω ότι δεν έχω πολλά να προσθέσω, γιατί εδώ επαναλαμβάνουμε μια συζήτηση που έχει ξαναγίνει και όλα όσα λέμε εδώ τώρα τα έχουμε ξαναπεί. Υπάρχουν εδώ δύο διαφορετικά ζητήματα το ένα είναι το περιεχόμενο μιας πολιτικής συμφωνίας και οι κανόνες εφαρμογής από εργασιακή, επιστημονική, ε, τεχνική, οικονομική σκοπιά. Και εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το ένα που έχει να κάνει με το περιεχόμενο της συμφωνίας και υπάρχει και το πολιτικό ζήτημα που αφορά τη Δυτική Σαχάρα. Και για αυτό το θέμα, όπως είπε και ο συνάδελφος Ρωμέβα, είναι πραγματικά ένα ζήτημα ξεκάθαρα πολιτικό, επομένως δεν είναι ουδέτερο. Οποιαδήποτε θέση ληφθεί για το θέμα αυτό δεν είναι μια θέση ουδέτερη, γιατί όλοι, όλοι εμείς γνωρίζουμε ότι για αυτό το θέμα υπάρχουν συγκεκριμένα συμφέροντα από την πλευρά του Μαρόκου και από την πλευρά της, Αργε... της της Αλγερίας και νομίζω ότι ο λαός της Δικής Σαχάρας για πάνω από 30 χρόνια ήταν αντικείμενο χρησιμοποίησης αυτών ε, των ε, συμφερόντων. Και λοιπόν ε, λυπάμαι πάρα πολύ που ε, υπάρχουν ε, κάποιες ευθύνες από την πλευρά του Μαρόκου που δεν έχει υλοποιηθεί αυτό το δημοψήφισμα για ε, που δεν είναι αρμόδιοι σε χρέο να αποφασίσουν για το μέλλον τους. Όμως τώρα εδώ αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι αν ωφελείται ή όχι ο πληθυσμός της Δυτικής Σαχάρας από αυτή τη συμφωνία. να απορρίψουμε τη συμφωνία σίγουρα δεν θα ωφεληθεί. Αν κρίνουμε τη συμφωνία θα πρέπει να μπορούμε να ελέγξουμε και να επαληθεύσουμε αν ωφελείται αυτός ο πληθυσμός συγκεκριμένα ή όχι. Γι' αυτό εγώ νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια κάπως παράδοξη κατάσταση Δηλαδή κάποιοι που λένε ότι υπερασπίζουν ε, τα συμφέροντα του λαού της Σαχάρας ε, απορρίπτουν αυτή τη συμφωνία. Και εγώ νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να αναλάβει κάθε πρωτοβουλία για να βρεθεί μια οριστική λύση για να μπορούμε να πιέσουμε για να γίνει αυτό το δημοψήφισμα όσο δυνατό πιο γρήγορα. Αλλά εγώ νομίζω ότι αυτό δεν είναι ασύμβατο με την έγκριση αυτής της συμφωνίας γιατί έτσι ως έχει μπορούμε να ελέγξουμε αν θα εφαρμοστεί σωστά και αν όχι θα μπορέσουμε να τερματίσουμε τη συμφωνία αυτή. Ευχαριστώ κύριε Κάπουλα, Ο κύριος Μιλάνα. Εγώ πιστεύω ότι η συζήτηση δεν θα πρέπει να οδηγηθεί προς το να λύσουμε εμείς ε, το πρόβλημα του λαού της Δυτικής ε, Σαχάρας. Γιατί ουσιαστικά θα είναι έτσι ένα όπλο για να προωθήσουμε ένα πολιτικό όπλο για να ξεκαθαρίσει η κατάσταση σε σχέση με το τι γίνεται σε αυτήν την περιοχή του κόσμου. Εμεί πριν ένα-δύο χρόνια απορρίψαμε μια συμφωνία. Το Κοινοβούλιο απέρριψε αυτή τη συμφωνία. Την ίδια ημέρα δόθηκε εντολή στην Κομισιόν με μια διαφορετική ψήφο από αυτή που είχαμε για την απόρριψη της συμφωνίας λέγοντας «Επιτροπή, εσύ πρέπει να ελέγξεις και να επαληθεύσεις μία σειρά ζητημάτων». Τώρα, και η δεύτερη ψήφος έχει ισχύ και η δεύτερη έχει ισχύ. Και η πρώτη έχει ισχύ και η δεύτερη έχουν ισχύ. Τώρα, εμείς στην δεύτερη περίπτωση ήμασταν απόλυτα ικανοποιημένοι. Δεν υπάρχει πλέον πρόβλημα συμβατότητας, ε, περιβαλλοντικού χαρακτήρα, δεν υπάρχει πρόβλημα περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, δεν ε, συνδέεται το θέμα το ισοβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην τελευταία γραμμή της συμφωνία. Δεν υπάρχει δυνατότητα αναστολής αυτής της συμφωνίας. Εγώ πιστεύω ότι η ψήφο του Κοινοβουλίου οδήγησε την Κομισιόν στο αναγκαστή να κάνει μια καλή συμφωνία, καλύτερη από αυτή που μας παρουσίασαν στο παρελθόν. Τώρα, αν εμείς δεν το λάβουμε υπόψη αυτό, δεν θα μπορέσουμε να βγούμε από αυτή την κατάσταση, γιατί διαφορετικά η προσέγγιση είναι ιδεολογική. Και στην Επιτροπή Αλίας δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή την ιδεολογική αντιπαράθεση που είναι ένα μικρό κομματάκι όλη τη σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Μαρόκο. Υπάρχουν και άλλα συμφέροντα αν θέλουμε να τα χτυπήσουμε στη σχέση Μαρόκο-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, ποιο είναι το ζήτημα πολιτικό κατά την άποψή μου. Ναι, αυτό είναι το ισχυρό πολιτικό ζήτημα. Είναι ότι αυτή τη φορά πρέπει να κάνουμε το αντίθετο από αυτό που κάναμε στο παρελθόν. Δηλαδή ακριβώς το αντίθετο. Να δράσουμε έτσι ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Ευρωπαϊκά Όργανα στο σύνολό του να αντιμετωπίσουν το μαροκινό ζήτημα. Αυτή τη φορά πρέπει να πούμε ναι λοιπόν στη συμφωνία, αλλά να πούμε και ναι στο γεγονό ότι το Κοινοβουλίο θα δείξει στην Κομισιόν το δρόμο να σκίσει πολιτική και στο ΝΟΙΕ να υπάρχει ένα ενεργό ρόλο εξωτερική πολιτική από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ερνούμε εγώ τώρα στην Επιτροπή Ελία εδώ να μπορούμε να, να είναι ο τόπο όπου θα πρέπει να καθορίζουμε την εξωτερική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ νομίζω ότι η συνάδελφος Φράγκα έχει συντάξει μια πολύ καλή γνωμοδότηση. Πιστεύω ότι η συμφωνία είναι καλή συμφωνία για τα θέματα που άπτονται τη Αλίας. Όμως όλο αυτό το θέμα νομίζω ότι θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε για να υψώσουμε τους τόνους έτσι ώστε η πρόταση που θα φτάσει στο Κοινοβούλιο να είναι ισχυρή για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της Δυτικής Σαχάρας. Διαφορετικά εμείς πάλι θα ξανακάνουμε το ίδιο λάθος, θα διαιρέσουμε το Κοινοβούλιο μεταξύ αυτών που θέλουν και που δεν θέλουν και κάποιοι θα συνδέονται με ορισμένα επιχειρήματα κάποιοι με κάποια άλλα και το θέμα τελικά της Δυτικής Σαχάρας ποτέ δεν θα αντιμετωπιστεί. Η πρόταση που πρέπει να υποστηρίξουμε είναι να καταλήξουμε σε μια συμφωνία για να έχουμε πράξεις, όχι απραξία. Δηλαδή, τώρα αν ε, το αποτέλεσμα θα είναι ε, απλά να έχουμε ένα χειροκρότημα στο τέλος, τελικά δεν θα έχουμε αντιμετωπίσει ούτε το πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Αλίας, ούτε το πρόβλημα του λαού της Δυτικής Σαχάρας. Ευχαριστώ κυρία Μιλάνα. Νομίζω ότι είχαμε μια ευρύτατη συζήτηση. Και θα ολοκληρώσουμε, θα έλεγα τώρα, να δώσουμε καταρχήν το λόγο στην Κομισιόν πως θέλει να διευκρινίσει κάποια ζητήματα και κατόπιν θα ξαναδώσουμε το λόγο στην συγγήτρια. Κύριε Ντεπίπερ. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Λόγω της ποιότητας της συζητήσεως δεν θα επαναλάβω πολλά από τα επιχειρήματα τα οποία εκφράστηκαν, εντυπωσιάστηκα. Απλώς μερικά σημεία. Πρώτον, ως διαπραγματευτές τηρήσαμε την εντολή και όλες τις συστάσεις που μας δόθηκαν. Αυτό προκύπτει από το ψήφισμα. Παρουσιάσαμε ένα πρωτόκολλο που ανταποκρίνεται ε, με τα όσα ζήτησε αυτό το Κοινοβούλιο. Ένα θέμα τέθηκε σχετικά με την αξιολόγηση των αποθεμάτων, ε, των πλεονασμάτων, των αλλιευτικών Νομίζω κάτσαμε με τους επιστήμονες του Μαρόκου, κάναμε αυτή την ανάλυση και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα βιωσιμότητας ως προς το θέμα αυτό. Επιπλέον, σε σχέση με το σχόλιο του κυρίου Μιλάνου που είναι πάρα πολύ εύστοχο και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα έχουμε τα μέσα για να παρακολουθήσουμε την εκτέλεση αυτού του πρωτοκόλου. Αν δεν υπάρχει αλία, δεν μπορεί να υπάρξει περιφερειακή ανάπτυξη αν δεν έχουμε τέτοιο πρωτόκολλο. Αν δεν υπάρχει αλίευση, άλλοι θα αλιεύουν και αυτό το οποίο έχουμε ως δυνατότητα να παρακολουθήσουμε την ανάπτυξη των ε, δραστηριοτήτων, τότε τι θα γίνει. Και αν δεν υπάρχει αλία, δεν θα υπάρχει καμία παραγωγικότητα. Έχουμε ε, τους μηχανισμούς εδώ για να εποπτεύσουμε την περιοχή. Έχουμε τα πρακτικά εργαλεία για το σκοπό αυτό. Για τα υπόλοιπα δεν χρειάζεται να προσθέσω οτιδήποτε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Φράγα για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ εξάγω τα εξή συμπεράσματα από τη συζήτηση. Το πρωτόκολλο που ήταν αντικείμενο διαπραγμάτευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σέβεται τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί και από αυτό το Κοινοβούλιο αλλά και από την εντολή του Συμβουλίου και από τη σκοπιά την κλαδική, της αλίας δηλαδή, σέβεται όλα όσα είχαν ζητηθεί. Είναι σύμμορφο όμως είχαν ζητηθεί. Επομένως, ε, βελτιώνει την κατάσταση σε σχέση με όλα όσα είχαμε στο προηγούμενο πρωτόκολλο, όμως οι μόνες ε, κριτικές που θα μπορούσαν να σταθούν και αναφέρομαι και σε γνώματα της άλλες επιτροπές, βασίζονται σε στοιχεία που τελικά έγιναν βάσει του προηγούμενου πρωτοκόλλου, που μόλις δεν ισχύουν για την ανάλυση αυτού εδώ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ωφέλη στον τοπικό πληθυσμό, για πρώτη φορά αυτό το πρωτόκολλο έχει τα κατάλληλα μέσα και θα γίνεται ένας έλεγχος εκ των υστέρων και έτσι θα δούμε αν λειτουργεί ή όχι. Και επομένω αν δεν λειτουργεί σημαίνει ότι θα ληφθούν τα μέτρα που έχουν προβλεφθεί για την αναστολή της συμφωνίας και την πάυση των πληρωμών. Από πολιτική σκοπιά θα ήταν πολύ εύκολο να πούμε ότι με μια θετική ή αρνητική θέση σε σχέση με το πρωτόκολλο θα λύνουμε το πρόβλημα της Δυτικής Σαχάρας. Όμως δυστυχώς δεν είναι έτσι. Εμείς δεν πρόκειται να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα της Δυτικής Σαχάρας είτε υπερψηφίσουμε είτε καταψηφίσουμε τη συμφωνία αυτή. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι το πολιτικό θέμα της Σαχαράς πάντοτε ανακύπτει όταν ε, μιλάμε για την Αλία που είναι ο πλέον αδύναμος κρίκος ε, στις σχέσεις μας με το Μαρόκο και ακριβώς ε, δεν προκύπτει, δεν ανακύπτει όταν μιλάμε για ένα προηγουμένο καθεστώς, ένα προνομιακό καθεστώς και επομένως εγώ νομίζω ότι το πολιτικό θέμα δεν πρόκειται να το επιλύσουμε εμείς. Υπάρχουν άλλα αρμόδια όργανα, ο καθένας μπορεί να έχει τη γνώμη του. Έτσι λοιπόν εγώ λέω ότι αυτή η συμφωνία είναι νόμιμη, και θα πρέπει να ελέγξουμε την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας. Εγώ θέλω και το Κοινοβούλιο να εμπλακεί περισσότερο στις Μικτές Επιτροπές, όπως σας είπα, έτσι ώστε όλοι να ενημερώνονται πλήρως για το τι συμβαίνει. Και εγώ πιστεύω λοιπόν ότι αυτή η συμφωνία είναι καλή. Νομίζω ότι έχει καταβληθεί μια σημαντική προσπάθεια στις διαπραγματεύσεις και πολλές από τις κριτικές που ακούσαμε εδώ από ορισμένου συναδέλφους θα ήθελα να έχουν γίνει και στη συμφωνία με τη Μαυριτανία, όπου δεν υπήρχε ούτε καν η ίδια διαφάνεια, ούτε η ίδια αυστηρότητα που είχαμε στην περίπτωση της συμφωνίας με το Μαρόκο. Πρόεδρο, ευχαριστώ κυρία Φράγα. Ολοκληρώθηκε και η συζήτηση. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών στις 6 Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Και περνάμε στο σημείο 11. Χρηματοοικονομική διαχείριση για ορισμένα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρέ δυσκολίε ε, ω προ τη χρηματοοικονομική του σταθερότητα. Η κυρία Πατράου είναι η συγγήτρια και τώρα θα έχουμε την πρόταση, την παρουσίαση της πρότασης από την Κομισιόν και θα κάνουμε και μία πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Παρακαλώ. welcome for your first time to the front of the Fisheries Committee? No, it's the second. Second? yeah. Oh, you were. Remember? Adelante, señor Oui, merci, monsieur le président. Excuse... Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Με συγχωρείτε. Σιωπή, παρακαλώ, λίγο ησυχία. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σας παρακαλώ, γιατί διαφορετικά θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Συνεπώς, θα σας παρουσιάσω αυτή την πρόταση ε, τροποποίησης ε, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλίας που είναι το top-up, τα πρόσθετα κονδύλια, όχι τα πρόσθετα κονδύλια, με συγχωρείτε, τις πρόσθετες καταβολές, ούτω ώστε τα κράτη-μέλη που έχουν δυσκολίες χρηματοδοτικές να προχωρήσουν με την εφαρμογή του προγράμματος του Ταμείου. Όπως ξέρετε, η κρίση οικονομική και η χρηματοπιστωτική των δύο τελευταίων ετών προκάλεσε δυσκολίες για ορισμένα κράτη-μέλη, αφενός επειδή το τραπεζικό σύστημα που έχει επηρεαστεί πολύ από την κρίση, την οικονομική και την χρηματοπιστωτική, διστάζει να συγχρηματοδοτήσει προγράμματα και έργα που τα κράτη-μέλη θέλουν να προωθήσουν στον τομέα της αλίας, της αντοτοκαλλιέργειας και της ανάπτυξης των παράκτιων ζωνών. Αυτές οι δυσκολίες του τραπεζικού συστήματος δυστυχώς συνδυάζονται με δυσκολίες ρευστότητα ε, των εθνικών ή τοπικών περιφερειακών διοικήσεων σε πολλά κράτη-μέλη, κράτη-μέλη που είναι τα κράτη-μέλη που είναι ε, υπό βοήθεια, που βοηθούνται ε, με ορισμένα μέσα οικονομικά που έχουν θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Επίτροπη πρότεινε ήδη εδώ και μερικά χρόνια το 2012 να θεσπίσει ένα σύστημα συμπληρωματικής χρηματοδότησης, ούτως ώστε τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να προχωρήσουν το συντομότερο δυνατόν με την εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται με την βοήθεια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλίας. ο κανονισμός που είχε υιοθετηθεί τότε έλυγε στις 31 Δεκεμβρίου 2013, διότι δεν ξέραμε ποιο θα ήταν το σύστημα που επρόκειτο να υπερισχύσει στη νέα περίοδο προγραμματισμού 2014-2020. Βλέπουμε τώρα ότι ο νέος μηχανισμός χρηματικής βοήθειας για την περίοδο 2014-2020 ανανεώνει το σύστημα αυτό βοήθειας προς τις χώρες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα. Η Κομισιόν λοιπόν βρίσκεται στην κατάσταση όπου είχε προτείνει και είχε υιοθετηθεί από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ένα σύστημα ενίσχυσης μέχρι το 2013 και θα έχουμε ένα νέο σύστημα που θα θεσπιστεί και θα παρατείνει την κατάσταση. Αλλά σχετικά με τα κονδύλια του Ταμείου, εάν δεν τροποποιήσουμε και πάλι τον κανονισμό του Ταμείου, όλα θα σταματήσουν στις 31 Δεκεμβρίου του 2013, πράγμα που θα είναι αν όχι παράλογο τουλάχιστον ε, περίεργο διότι θα έχουμε ένα σύστημα που θα σταματήσει το 2013 και ένα άλλο που θα αρχίσει αλλά το σύστημα του 2013 δεν θα μπορέσει να συνεχιστεί ούτε ακόμα και για τα προγράμματα που τρέχουν. Γι' αυτό προτείναμε αυτήν την τροποποίηση του κανονισμού που είναι απλή και που συνίσταται απλώς σε μια κατάργηση ενός άρθρου που περιόριζε στην 31η Δεκεμβρίου 2013 το, το καταργούσε το μηχανισμό και προτείνει την, παράστα, την παράτασή του μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015. Θα με ρωτήσετε ποιες είναι οι χώρες που μπορούν να ωφεληθούν από αυτό το σύστημα. Υπήρχαν αρχικά 7 χώρες που μπορούσαν να ωφεληθούν, αλλά όλες ε, δεν ζήτησαν να ωφεληθούν από το σύστημα αυτό. Οι χώρες που το αποφάσισαν και που ωφελήθηκαν και που θα μπορούσαν συνεπώς να ωφεληθούν από την παράταση του συστήματος αυτού είναι η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, όχι, όχι, όχι η Ρουμανία και η Κύπρος. Η Ρουμανία μπορούσε να ωφεληθεί, ναι, ναι, και η Ρουμανία, με συγχωρείτε, έκανα λάθος. Οι χώρες που μπορούσαν να ωφεληθούν και που δεν ωφελήθηκαν είναι η Λετωνία, η Ουγγαρία και η Ιρλανδία. Πρόκειται λοιπόν χωρίς καμία αύξηση των αρχικών πόρων που είχαν δοθεί στα κράτη-μέλη θα πρέπει να επιτρέψουμε στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία, στην Ρουμανία και στην Κύπρο να εξακολουθήσουν να υλοποιούν τα υπηρεσιακά προγράμματα του Ταμείου μέχρι τέλους 2015, εποφελούμενα από το σύστημα αυτό. Αυτή είναι η κατάσταση. Απλά πράγματα. Κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πατράου Νέβες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ νομίζω ότι ήδη η Κομισιόν μας παρουσίασε το πλαίσιο της έκθεσης αυτής και γι' αυτό θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω την Κομισιόν για αυτή την πρότασή της η οποία πραγματικά αποδίδει δικαιοσύνη. Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι υπάρχουν χρηματοοικονομικές, οικονομικές, κοινωνικές δυσκολίες σε γενικευμένο βαθμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα σε χώρες που είναι σε πρόγραμμα εξωτερικής βοήθειας όπως αυτές που, που αναφέρθηκαν και θα ήταν πραγματικά λυπηρό να προστίθονται και άλλες δυσκολίες που θα ποινικοποιούσαν σημαντικούς κλάδους όπως είναι ο κλάδος της αλίας. Άλλωστε, οι χώρες που αναφέρθηκαν πραγματικά έχουν πάρα πολύ ισχυρά συμφέροντα στον τομέα της αλίας και η κατάσταση στην οποία βρίσκονται θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τα επιχειρησιακά τους προγράμματα καθώς ε, θα οδηγούσαν και στην αύξηση των δυσκολιών σε σύγκριση με το τι συμβαίνει σήμερα. Επομένως, ε, με μεγάλη ικανοποίηση χαιρετίζω αυτή την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπογραμμίζεται ότι εδώ δεν πρόκειται για καμία αύξηση ε, άχθους για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν υπάρχει καμία αύξηση των ε, αξιών και των ε, κονδυλίων που θα δοθούν. Ο προπολογισμό παραμένει ο ίδιος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το τονίσουμε, γιατί υπάρχουν ε, συγκεκριμένες χώρες δικαιούχοι και κανένα κράτος δεν θα ζημιωθεί γιατί διατηρείται το ίδιο ανώτατο όριο στον προϋπολογισμό. Εδώ απλώς μιλάμε για να καταβληθούν, να μπορέσουμε να καταβάλουμε νωρίτερα κάποιες πληρωμές. Δηλαδή να δημιουργήσουμε μία πρόσθετη ευελιξία στο πρόγραμμα αυτό και εμείς πάντοτε μιλούσαμε για την αναγκαιότητα της ευελιξίας γιατί είναι αλήθεια ότι αν έχουμε 28 κράτη-μέλη από μία ένωση, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και σημαντικές διαφορές μεταξύ αυτών των κρατών μελών. Και πρέπει να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την ποικιλομορφία. Και πραγματικά αυτή η πρόταση της Κομισιόν λαμβάνει υπόψη την ποικιλομορφία. Και είναι πολύ σημαντικό να προσθέσω πως ε, σεβόμαστε εδώ την αρχή της επικουρικότητας προτείνοντας ένα μηχανισμό που επιτρέπει στην Κομισιόν να δώσει περισσότερη στήριξη στα κράτη που βρίσκονται υπό καθεστώς εξωτερικής βοήθειας Επίσης, ε, σέβεται την αρχή της αναλογικότητας, ε, καθώς ε, η παράταση του ποσοστού της χρηματοδότησης με αύξηση 10% λαμβάνει υπόψη και τις οικονομικές δυσκολίες και την οικονομική κατάσταση που βιώνουν τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή η πρόταση επίσης είναι ε, επιτακτικό να τεθεί σε εφαρμογή γιατί αυτή η προσάυξηση του 10% έχει διασφαλιστεί μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 2013 και επομένως εδώ πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχει διακοπή αυτού του μηχανισμού. Επομένως, ε, οι λέξεις αλληλεγγύη και απλούστευση αρμόζουν και στην περίπτωση αυτή στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και θα ήθελα να προσθέσω κάτι που νομίζω ότι δεν αναφέρθηκε από την πλευρά της Κομισιόν. Ότι είναι πάρα πολύ δίκαιο να προχωρήσουμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Λίας με τον ίδιο τρόπο που προβλέπεται να προχωρήσουμε και με τα άλλα ταμεία. Εμείς ε, ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή Υπάρχει ένας κανονισμός για το 2014-2010 που προβλέπει να εφαρμοστεί ένα top-up σε σχέση με όλα τα ταμεία και για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και που εμείς ψηφίσαμε πριν 10 μέρες περίπου. Προβλέπεται λοιπόν ένα top-up για όλα αυτά τα ταμεία μέχρι 30 Ιουνίου 2016 και επομένως δεν θα ήταν κατανοητό το ίδιο να μην γίνει με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλίας. Θα ήταν πραγματικά άδικο διαφορετικό γι' αυτό αυτή η πρόταση είναι απαραίτητη για να τύχει ίσης μεταχείρισης το ΦΕΠ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ελίας, σε σχέση και με όλα τα άλλα ταμεία που έχουν αντεχθεί στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020. Και το γεγονός ότι θα εφαρμοστεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016 σημαίνει ότι αυτό το top θα εφαρμοστεί και σε όλες τις δαπάνες που θα έχουν πληρωθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλίας. Δηλαδή, δεν θα μπορούσαμε εδώ να μην ε, λάβουμε υπόψη την πρόθεση της ε, Κομισιόν ε, όταν ίδρυσε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλίας. Αυτή είναι η πρόθεση της Κομισιόν για όλα τα άλλα ταμεία μέσα στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Και το ίδιο λοιπόν θα πρέπει να γίνει και για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλίας για να έχουμε ίση μεταχείριση για όλα τα ταμεία. Δηλαδή όχι μόνο παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016, αλλά επίσης και να λάβουμε υπόψη ότι όλες οι δαπάνες που θα καταβληθούν από το ΦΕΠ θα καλύπτονται από αυτή την αναθεώρηση του κανονισμού. Ευχαριστώ και πάλι την Κομισιόν για την πρωτοβουλία της, η οποία εν αυτό το χρόνο μπόρεσε να βρει μία λύση πάρα πολύ δίκαιη. Και εμείς ε, φυσικά θα προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε αυτό το χρόνο για να επιλύσουμε και αυτή την κατάσταση. Ευχαριστώ. Ε, Κανείς δεν μου έχει ζητήσει το λόγο. Επομένως, θεωρώ ότι ολοκληρώσαμε και αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων για το ζήτημα αυτό. Δεν υπάρχει προθεσμία τροπολογιών ακόμη. Είχαμε μόνο ανταλλαγή απόψεων. Μια ερώτηση. Θα πρέπει να περάσουμε στο επόμενο σημείο τη μερικής διάταξη που είναι το 13. Είναι αλήθεια ότι στις ψηφοφορίες που πάντα τις κάνουμε στην αρχή δεν ε, βάζουμε ώρα και είναι αλήθεια ότι υποχρεούνται οι βουλευτέ να παρευρίσκονται στην Επιτροπή τους και η ίδια η Επιτροπή μπορεί να αλλάξει την ημερησία διάταξη. Είναι σίγουρο ότι βέβαια στην ημερήσια δίταξη έλεγε εδώ ότι οι ψηφοφορίες θα γίνουν στις 6 παρατέταρτο. Τώρα, ε, με την επιφύλαξη ότι η Επιτροπή μπορεί να αλλάξει την ημερήσια διάταξη και ότι οι βουλευτές θα έπρεπε να παρευρίσκονται εδώ, εγώ θα πρότεινα να κάνουμε ένα διάλειμμα 10-15 λεπτά και να αρχίσουμε. Το λάθος που κάναμε είναι ότι βάλαμε ώρα εδώ. Αν και βέβαια, όπως σας είπα, υποχρεούνται οι βουλευτές να είναι στην Επιτροπή τους. Αλλά τέλος πάντων κάπως έλεγε εδώ στο σχέδιο της ημερησίας διάταξης ότι θα ψηφίσουμε στις 6 παρατέταρτο, πως κάποιος δεν ήρθε ακόμη. Επειδή πιστεύει ότι τότε θα γίνουν ψηφοφορίες. Σας κάνουμε ένα διάλειμμα και θα αρχίσουμε τις ψηφοφορίες ακριβώς στις 6 παρατέταρτο. Έχουμε μια μακρά ψηφοφορία και πάμε. Θα διακόψουμε για 15 λεπτά.

Vayan tomando asiento. Take your seats, please. Καθίστε παρακαλώ. Je Είστε έτοιμοι, ωραία. Να ξεκινήσουμε με το σημείο 13 και την ψηφοφορία της έκθεσης Αρσένη. Θα το κάνουμε ηλεκτρονικά, αν και υπάρχουν πολλές συμβαστικές, αλλά εγώ νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και νομίζω ότι θα πάρει λιγότερο χρόνο. Αν ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, έχετε όλοι τι κάρτε σα. Είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε. Λοιπόν, υπαριθμόν 8 συμβαστική τροπολογία. Πέρας. Δεν φάνηκε να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα. Να ξαναρχίσουμε. Εντάξει. Ουλριχ. Ψηφίζουμε τη συμβαστική 8. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία. 150. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 153. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 154. Άρχεται τη ψηφοφορία. Τέλος. 154. Ξαναρχίζουμε. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 155. Αρχή. Λέξη. Απορρίπτεται. Συμβαστική 9. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 18. Στη σελίδα 7 λέει ο πρόεδρος. Τροπολογία 18.

Τροπολογία 182. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 19. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 10. Ε, αρχή. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβασμός 12. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Θεροπολογία 209. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβασμός 13. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 37. Σελίδες 25-26 λέει ο πρόεδρος. Τροπολογία 37. Τη βρήκατε. Αρχή. 25-26 σελίδα. Τροπολογία 37. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 38. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 39. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 15 αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 261. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτει. Συμβαστική 16. Ποιοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 46. Στα σελίδα 32 ή 33. 46. Υπέρ. Αρχή μάλλον, με συγχωρείτε. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία. 274. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 17. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στη σελίδα 36 και 37. 295 τροπολογία. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Νίξο Καντέκ. 296. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 62. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 63. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 64. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 65. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 66. Αρχή. Απορρίπτεται. Συμβασμό 18. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 300. Εκεί. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 19. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 305. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβασμός 20. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 311. Αρχή. επί 11. Να κλείσουμε. Απορρίπτεται. 78. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Ένφυση 47. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 313. Αρχή. Πέρας. Αγκρίνεται. Συμβεσμός 21. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβασμός 22. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβασμός 23. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Πάμε στη σελίδα 46-47, τροπολογία 90. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 92. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 91. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Envy. Όχι. NV1. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 94. Αρχή. Εν Εγκρίνεται. δύο. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβεσμός 1. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 96. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Εκατόν δύο. 102. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβασμός 2. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 104. Αρχή. Πέρας. Μπορείτε. Τροπολογία 105. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Τερπολογία 106. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 107. Αρχή. Πέρας τον οκτώ. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 109. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 113. έχει Πέρας. Απορρίπτεται. 114. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 115. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβασμός 3. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 123. Και είναι ταυτόσιμη με τις 124 και 125. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβασμός 4. Αρχή. Συμβασμός 4. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 132. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 133. Αρχή. Πέρας. Ρετσαθάδα. Απορρίπτεται. Συμβασμός 5. Υπέρ. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 6. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 7. Άρχη την ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 141 που είναι ταυτόσιμο με την nv Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 142 αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 144. Αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 145, ταυτόσημη με την 146 και την nv αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. 147 αρχή. Πέρας. Απορρίπτεται. Να περάσουμε στη νομοθετική πρόταση όπως τροποποιήθηκε. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται 19 υπέρ, καμία ψήφος κατά, 4 αποχές. Και πρόταση ψηφίσματος όπως τροποποιήθηκε, ψηφίζουμε στο συνολό της αρχή. Γκρίνεται. Με το ίδιο αποτέλεσμα. Συγχαρητήρια κύριε Αρσένη. Sí, señor Arsenis. Just. Thank you, President. Colleagues, I know that this was a very, very long. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ξέρω ότι ήταν μακρύς ο δρόμος μας. Στην έκθεση αυτή υπάρχουν πράγματα που αρέσουν ε, σε κάποιους ε, και δεν αρέσουν ε, σε κάποιους. Δηλαδή όλοι βρίσκουν κάτι που τους αρέσει και που δεν τους αρέσει. Έτσι είναι η δημοκρατία. Καταφέραμε να βρούμε κοινό τόπο εντός της Επιτροπής μας και νομίζω ότι αυτό αξίζει να το γιορτάσουμε. Ήρθαμε από πολύ διαφορετικές κατευθύνσει και καταφέραμε να βρούμε πλειοψηφία μια πρόταση που βρήκε την υποστήριξη της πλειοψηφίας στο θέμα αυτό και ε, θα ήθελα να καλέσω τους ε, συναδέρφους ε, στο μπαρ Mickey Mouse σε λίγο για να γιορτάσουμε. Νομίζω ότι πρέπει να γιορτάσουμε τη δημοκρατική διαδικασία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Αρσένη. Συχνά επικρίνω την Επιτροπή μας και θα ήθελα, αλλά θα ήθελα να ε, σας επενέσω που ε, προχωρήσατε το θέμα αυτό και μάλιστα στο, στο σωστό ρυθμό. Ίσως κάποιοι αντιπρόεδροι στην ε, Ολομέλεια να μπορέσουν να ακολουθήσουν το παράδειγμά σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και καθώς προέρχεται από εσά αυτό, το, το εκτιμώ ακόμη περισσότερο. Δεν έχουμε τίποτα στα διάφορα. 15 στην ημερομηνία τη επόμενη συνεδρία, 27 Νοεμβρίου και το πρωί και το απόγευμα και στι 28 μόνο το πρωί. Ευχαριστώ όλου και ολοκληρώνεται η συνεδρίασή μα.